So, Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε 9 και 6 λεπτά. 6 ε, λεπτά καθυστέρηση, δεν το συνηθίζω. Αλλά μια και δεν είμαστε και πολύ αριθμοί. Θα αρχίσω πιο αργά πριν ξεκινήσουμε τις εργασίες μας, θα δώσω το λόγο στους διερμηνείς για να κάνουμε μια ανακοίνωση. Οι διερμηνείς σας ενημερώνουν ότι έχουμε μπει στη 17η ε, ημέρα των κινητοποιήσεων και ότι ενώ ορισμένε καμπίνες μόνο έχουν επιταχθεί προκειμένου να μην τους επιτραπεί να γίνει απεργία, άλλες όπως η ελληνική δεν έχουν επιταχθεί. Εμείς σε ένδειξη αλληλεγγύη συνεχίζουμε την ε, συνεδρίαση, δεν διακόπτουμε, δεν κάνουμε στάση εργασία σε ένδειξη αλληλεγγύη προ του συναδέλφου μα. Ωστόσο, η συνεδρία θα σταματήσει ακριβώ στι 12.30. The exchange of views on the negotiation for a deep and comprehensive free trade agreement EU Tunisia. Περνάμε στην, ε, στο θέμα της ε, Συμφωνίας Ελεύθερων Αλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης Τινησία. Μετά την Αραβική Άνοιξη ε, ήταν πολύ σημαντικό να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στην Τινησία ε, η οποία ε, ε, είχε διαταραχθεί. Έχουμε πολλές επίσης οικονομικές εξελίξεις στην Τινησία. Μετά το δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων ε, που έγινε πριν από δύο-τρεις εβδομάδες που ήταν μάλιστα και πολλά υποσχόμενος ε, έχουμε μια καινούργια κατάσταση ελπίζω ε, ένα καινούργιο ορίζοντα από ευκαιρίες Εμείς ε, με την Κομισιόν έχουμε μια συμφωνία διαφάνειας Το πρωτόκολλο των πρακτικών της διαβρομάτευσης αυτής του δεύτερου γύρου θα δημοσιευθεί στο μισθότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Trade. Η συνεδρίασή μας έτσι κι αλλιώς ε, εκπέμπεται μέσω του ίντερνετ. Καλωσορίζω λοιπόν και όλο το απομακρυσμένο κοινό μας για να συζητήσουμε τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις. Έχουμε μαζί μας εμπειρογνώμονες από την Τινησία, Λομπράν Γερίμπη, που είναι η πρόεδρος της, του Σολίντα από την Τινησία, και ο κύριος Καρίμ Νταβούτ, τη Συναγκρή τη Ομοσπονδία Τινησίας, Την Ισία. Πριν του δώσω το λόγο, θέλω να καλωσορίσω την κυρία Μόνικα Χέντσκι, που είναι προϊστάμενη της μονάδας για τις ε, χώρες του Μαγκρέμπ. Από την πλευρά της Κομισιόν θα μας ενημερώσει ε, για τις απόψεις της Κομισιόν. Κυρία Γερίμπη, Οκτώ λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Λάγκε. Είμαι παλιότερη πρώην βουλευτής και πρόεδρος και ιδιωτικό μέλος της, ε, του ε, του Think Tank Solida που ασχολούμαστε με θέματα οικονομία, ε, ενέργεια κλπ. Από τον Νοέμβριο 2011 η Τινησία είναι ε, ε προνομιούχο εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η δημοκρατική μετάβαση έχει προχωρήσει. Ε, η συνέλευσή μας ε, είναι η συμμετοχή των γυναικών. Έχουμε δημοκρατικούς θεσμούς πλέον. Έχουμε ένα σχέδιο αποκέντρωσης. Η κοινωνικο-οικονομική όμως μετάβαση αντιμετωπίζει δυσκολίες εξαιτίας και ενδογενών αλλά και εξωγενών παραγόντων. Αυτοί οι παράγοντες ε, θέτουν σε κίνδυνο την ε, δημοκρατία. Γι' αυτό λόγο χρειάζεται να καθορίσουμε μια καινούργια εταιρική σχέση με Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ισίας με πάνω στην αρχή της ε, συνανάπτυξης, της παράλληλης ανάπτυξης. Ε, με ένα τρόπο που θα απορροφήσει τις, ε, μεγά, τη μεγάλη ανεργία των νέων και των διπλωματούχων. Χρειαζόμαστε επενδύσεις, ευρωπαϊκές επενδύσεις στην Τινησία έτσι ώστε η Τινησία να ανέβει στις διεθνείς ε, αλυσίδες αξίας για να αποφύγουμε κιόλας το brain drain, την μαζική αποχώρηση των επιστημόνων μας αλλά και όχι μόνο ε, πολλών ανθρώπων που ε, περνούν την Μεσόγειο προκειμένου να μεταναστεύσουν. Πριν σας μιλήσω για την ε, σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, να σας πω τι έχουμε κάνει από το Σεπτέμβριο 2015. Για μας αυτή η ζώνη ελεύθερων συναλλαγών πρέπει να δημιουργηθεί με διαφάνεια. Το 2016 προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε το κοινό μας, τους φορείς μας, απλοποιώντας τις διατάξεις της ε, συμφωνίας. Ε, επιμένουμε στην ανάγκη να γίνουν τομεακοί, κλαδικές τομεακές μελέτες και το 2018 ε, ξεκινήσαμε μια προσφορά σε συνεργασία με το Υπουργείο ε, τους φορείς ε, της κοινωνίας των πολιτών ε, για το θέμα των υπηρεσιών ε, πληροφορικής. Πάντοτε σε διάλογο με τα αντίστοιχα επαγγέλματα. Καταλήξαμε σε εξής συστάσεις. Πρώτον, χρειαζόμαστε μια ένα εκ των προτέρων όραμα πολιτικό και οικονομικό της καινούριας εταιρικής σχέσης που θα επιτρέψει στην στρατική, τη στρατηγική της παράλληλης ανάπτυξης. ψηφιακή μετάβαση, ενεργειακή μετάβαση, με καινούριε υποδομές και καλώδια για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών. Ε, τουρισμός, ε, logistics, ε, που πρέπει επίσης να αναπτυχθούν μαζί με τον τουρισμό, με τις μεταφορές για να στηριχθεί ο τουρισμός. Η προσέγγιση της ζώνης ελεύθερων αλλαγών πρέπει να είναι κλαδική, τομεακή, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους ε, των φορέων. Ε, από κάτω προς τα πάνω. Οι εκπρόσωποι των διαφόρων επαγγελμάτων θα πρέπει να διαμορφώσουν τη δική του στρατηγική. Ε, η ζώνη ελεύθερων συναλλαγών θα πρέπει να είναι ένα εργαλείο για την εφαρμογή της δικής μας τομεακής στρατηγικής κάθε φορά. και η Σολίντα και πολλοί εκπρόσωποι τη κοινωνία των πολιτών το υποστηρίζουν. Ε, Επίση, χρειαζόμαστε μια προσέγγιση με ε, θετικού καταλόγου. Μιλούμε για υπηρεσίε και εδώ έχουμε πολλέ διαφοροποιήσει. Χρειάζεται να έχουμε λοιπόν ένα κατάλογο και να διατηρήσουμε του ευαίσθητου και να προασπίσουμε του ευαίσθητου τομεί. Τέλος, συμμετοχική προσέγγιση με αποτελεσματική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. ε, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για μια συμφωνία. Μεταξύ αυτών η κινητικότητα των ατόμων. Ε, μην μπερδεύουμε την κινητικότητα με τη μετανάστευση. Είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για απελευθέρωση των υπηρεσιών, ε, για ίση συμμετοχή και πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά αν δεν εξασφαλιστεί η κινητικότητα και προφανώς η κινητικότητα των επαγγελματιών που είναι η κορονίδα ε, αυτής της διαδικασίας. Επίσης, σταδιακή προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τον ρυθμό της ε, Τινησίας, ε, μια που βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο, σε μια σχετική αστάθεια. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερο χρόνο. Ε, ισότητα στην πρόσβαση στις υπηρεσίες και στη χρηματοδότηση, στα ταμεία, πολύ σημαντικό θέμα αυτό, στήριξη της ε, σαν αν, αμοιβαία αναγνώριση των ε, διπλωμάτων. Ε, μιλάμε επίσης για ε, κανονιστική σύγκληση. πιστεύουμε ότι εκεί θα πρέπει και η Τινσία να έχει φωνή. Δυστυχώς όμως δεν εκπροσωπούμαστε στην νομοθετική διαδικασία και στα νομοθετικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε χρειάζεται να εξετάσουμε μια ενδεχόμενη συμμετοχή της Τινησίας στα όργανα που νομοθετούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δίνουμε τη γνώμη μας, για να ε, γίνεται μια διαβούλευση ε, εν ώψη οποιοδήποτε νομοθετικού κειμένου εγγράφου που θα μας ε, επηρεάζει πρέπει να διατηρήσουμε το δικαίωμά μας ε, να αριθμίζουμε την αγορά μας μέσω της ε, ε, ζώνης ελεύθερων συναλλαγών και να μην είμαστε πλέον υποψήφοι στους ε, καταλόγους, στον κρύο και το μαύρο κατάλογο, όπως και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν έχουμε μια τέτοιου είδους συμφωνία, δεν είναι δυνατόν ταυτόχρονα να είμαστε και υποψήφοι στο, για το μαύρο και τον κρύο κατάλογο. Οι συμφωνίες και τα κεφάλαια αυτή τη στιγμή ως έχουν είναι ασύμετρα. Ασύμετρα υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο πολύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα είχε συμφέρον να ενισχύσει τους εταίρους της ε, για μα, η ε, σφαιρική και σε βάθο ζώνη αίθουσα Αναλλαγών, είναι μια, ένα εργαλείο προκειμένου να φτάσουμε σε ένα καινούριο κοινωνικό-οικονομικό μοντέλο που θα ικανοποιεί τις φιλοδοξίες μα. Ε, δύο προβλήματα έχουμε. Ε, οι, περιφερειακές, οι διαφορές μεταξύ ε, ανάμεσα στι περιφέρειέ μα και η ανεργία των νέων και των διπλωματούχων μα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια καινούργια εταιρική σχέση που θα είναι ιδιαίτερη, προνομιακή και θα λαμβάνει υπόψη το ότι η Τινησία βρίσκεται σε δημοκρατική μετάβαση. Ευχαριστώ. In time. Απολύτως και στην ώρα σας ακριβώς και με σαφές μήνυμα. Κάριμ Νταούτ, παρακαλώ, από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γεωργίας. Έχετε το λόγο. την συγγνώμη. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα ε, τελευταία δύο χρόνια η γεωργία της Τινησίας έχει πραγματοποιήσει σημαντικές πρόοδους, εξασφαλίζοντας αυτάρκεια σε αρκετά προϊόντα, γάλα, οποροκυπευτικά και έτσι περιορίζοντας την εξάρτηση από τις ε, εισαγωγές, αλλά και βελτιώνοντας τις εξαγωγικές της αγορές. Ωστόσο, ο μιλητής διαβάζει ένα κείμενο το οποίο δεν μεταφράζεται στην ταχύτητα στην οποία το αναγνώσκει πρέπει να διερωτηθούμε τι είδους γεωργία μπορούμε να ετοιμάσουμε και αν μπορούμε να θρέψουμε όλους τους ανθρώπους. Η γεωργία της Τινησίας έχει φτάσει σε επίπεδα μεγάλης ποικιλία και βελτίωσης του κόστους παραγωγής με όλες τις απειλές της κλιματικής αλλαγής και την ευαισθητοποίηση. Ο ομιλητής δεν πρόκειται να μεταφραστεί στο ρυθμό στον οποίο αναγυγνώσει και το κείμενό του. Υποφέρει λοιπόν από μείωση του μεριδίου στην ΑΕΠ, στο ΑΕΠ, ο τομέας της γεωργίας, έχει μεγάλη ε, ποικιλία, αντιμετωπίζει τις απειλές της κλιματικής αλλαγής, της ε, σπάνιδας και της, ε, του εύθραυστου των φυσικών πόρων. Δεν έχει ικανοποιητική οργάνωση της αλυσίδας παραγωγής και διάθεσης του κόσμου της γεωργίας, δεν είναι ελκυστικός για τους νέους και επίσης υπάρχουν και προβλήματα διακυβέρνησης, ε, θεσμικής υποστήριξης, πολιτικού οράματος. Οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις είναι μεγάλη. Και βέβαια ταυτόχρονα έχουμε την απελευθέρωση των εμπορικών μας ε, συναλλαγών και ιδιαίτερα αυτών με τους Ευρωπαίους εταίρους στο πλαίσιο της ΑΛΕΚΑ. Για να αντιμετωπιστούν λοιπόν αυτοί οι κίνδυνοι, και αυτές οι προκλήσεις, χρειάζεται μια καινοτόμα και θαραλέα προσέγγιση για την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα. Από το 2011, την Επανάσταση στην νησία και το Δημοκρατικό Άνοιγμα και τον συνδικαλιστικό πλουραλισμό δημιουργήθηκε η Συνάγκρη, το συνδικάτο μας. Ωστόσο, ακόμα χρειάζεται πολύ μεγάλη ε, προσπάθεια για την βελτίωση της αποδοχής του. Πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε 80% των γεωργών της Τινησίας με λιγότερο από 10 εκτάρια. 70% από αυτούς έχουν λιγότερα από 5. 80% των κτηνοτρόφων βοηδών έχουν λιγότερο από, λιγότερες από 10 αγελάδες και 70% από αυτούς λιγότερες από 5. Αλλά αυτή η μικρή κλίμακας γεωργία καλύπτει το 70% της συνολικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων στην Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια προσπάθεια να αναπτύξουμε και τα συστήματα της άρδευσης και την αξιοποίηση των όμβριων υδάτων και την αλυσίδα αξίας, τη, τη βιολογική γεωργία, τις ενδείξεις προελεύσεως, την μεσογειακή διατροφή και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η γεωργία στην Τινησία με συνεταιρισμούς που ακόμα δεν έχουν αναπτυχθεί στη χώρα μας ικανοποιητικά προς όφελος των μικρότερων γεωργών, εκείνων που ζουν σε λιγότερο ε, αποδοτικές γεωργικά περιοχές και βεβαίως πρέπει να αγωνιστούμε για οι διερμηνείς δεν πρόκειται να μεταφράσουν τον ομιλητή όταν διαβάζει το κείμενο στην ταχύτητα με την οποία το διαβάζει. Συνεχίζουμε με χαμηλές βροχοκοπτώσεις που για την περιοχή μας, το Μαγκρέμπ γενικότερα, οδηγεί σε απώλεια σημαντικού αριθμού των αρρώσιμων γεών η ξηρασία θα οδηγήσει σε απώλεια της ελαιοπαραγωγής και της κτηνοτροφίας των βοηδών. Πρέπει να ενισχύσουμε την πράσινη γεωργία και να βελτιώσουμε τις συνθήκες για τη γεωργία της Τινησίας, η οποία διαδραματίζει ρόλο κινητήριου μοχλού για την αντιμετώπιση των μεγάλων κρίσεων που αντιμετωπίσαμε και το 7 και το 11 και το 14. Έχει συμβάλει το μέγιστο στην ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια των κρίσεων αυτών, εξασφαλίζοντας την επιβίωση της οικονομίας της χώρας μας. Πρέπει να θεωρηθεί λοιπόν ως αποδοτική οικονομική δραστηριότητα αυτή η γεωργική, να μην υφίσταται τις πιέσεις με τον πληθωρισμό των τιμών που χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι του πληθωρισμού, να στηρίξουμε την βιώσιμη ανάπτυξη, να βελτιώσουμε την ισότητα πρόσβασης στις αρρώσιμες γεές, αλλά και στις αγορές, να εξασφαλίσουμε συστήματα ανθεκτικά γεωργικής παραγωγής, με βιοπικιλότητα, με γενετική ποικιλομορφία. Εμείς, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μιλούμε για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα πέραν των στενών οικονομικών συμφερόντων. Η την ίση γεωργή και αλληλείς περιμένουν τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση μας από το πρόβλημα αυτό ως ένα παράγοντα σταθεροποίησης και ανάπτυξης που θα είναι επωφελής και για σας, γιατί ο περιορισμός των ανισοτήτων μεταξύ των μοντέλων γεωργικής παραγωγής που έχουμε θα είναι επιζήμιος και για τις δύο πλευρές. Επομένως, τεχνικά, επιμελητιακά και άλλα οικονομικά μέσα που μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας επιτρέψουν να ανέβουμε επίπεδο μέσα στην επόμενη πέντα αιτία. Πρέπει να μιλήσουμε όχι μόνο για τα ευάλωτα προϊόντα, στη ε, συζήτηση για την αποδιάρθρωση του συστήματος τιμών εισόδου, γιατί μπορεί να είναι ανταγωνιστικά τα γεωργικά προϊόντα, αλλά χρησιμοποιούνται και ως φραγμή στην είσοδο της αγοράς. Έτσι λοιπόν μπορούμε χάρη στην ελπίδα αυτή, να, στην ε, συμφωνία αυτή να ελπίζουμε ότι μπορούμε να έχουμε μία πρόοδο με βάση και την ε, οικονομική συνεργασία που θα καθησυχάσει και θα ωφελήσει τους γεωργούς της Τινησίας και θα τους πείσει να συμμετάσχουν σε ένα εγχείρημα για το μέλλον. Η Ευρώπη πρέπει να δείξει θάρρος πολιτικό, πρέπει να στηρίξει τη γεωργία μας, όπως στήριξε τη γεωργία της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, για να έχουμε ένα χώρο ελευθερίας, εμπορίου, ανάπτυξης, εταιρικής σχέσης με ένα συνολικό σύστημα γερό, στεναρό, προς όφελος και των δύο πλευρών. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τεθεί σε εφαρμογή αυτή η συμφωνία. Την υποστηρίζει εννοείται το συνδικάτο μας την έχουμε αναπτύξει συνεργασία με την ε, Adenauer Conrad Stiftung και με άλλους φορείς και οργανώνουμε συζητήσεις τρογγυλής τραπέζης. Σε εθνικό επίπεδο επίσης αναπτύσσουμε τη δουλειά μας για να κοινοποιήσουμε την ε, συμφωνία αυτή σε όλους τους γεωργούς της Τινησίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα θέλαμε να ξέρουμε πόσο ισορροπημένη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στις διαπραγματεύσεις και πόσο προστατευμένος είναι ο γεωργικός κλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σε κάποια κράτη-μέλη. Μόνικα, έχεις το λόγο για πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και τους δύο προηγούμενους ομιλητέ, οι οποίοι νομίζω ότι παρουσιάζουν εδώ στο Κοινοβούλιο την άποψη της Κοινωνία των πολιτών στην ε, την Ισία. Θεωρώ ότι ήταν πολύ επιτυχή ο δεύτερο ε, γύρο στην Ισία πρόσφατα και ασφαλώ μια και πάντα συναντούμε εκπροσώπους της κοινωνία των πολιτών ε, πέρα από τους εκπροσώπους της Τινησιακή κυβέρνησης. Καλωσορίζουμε λοιπόν την διαφάνεια τη διαδικασία αυτή ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη δημοσίευση των ε, εγγράφων αυτών, γιατί πάντα τα δημοσιεύουμε. Υπήρχε λοιπόν δύο χρόνια καθυστέρηση μεταξύ του προηγούμενου γύρου διαπραγματεύσεων και του τωρινού γύρου διαπραγματεύσεων. αλλά και η κυβέρνηση, αλλά και η τυνησιακή πλευρά ήθελε να χρησιμοποιήσει όλο τον χρόνο που είχε για να είναι σίγουρη για τη διαδικασία. Αυτό για να σας δείξουμε την ε, διαφάνεια στην διαδικασία αυτή. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτά που είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητέ, σε ό,τι αφορά δηλαδή την ανάγκη να υπάρχει ε, ανάγκη για να υπάρχει διαφάνεια. Η ΑΛΕΚΑ φυσικά δεν είναι μια οργάνωση η οποία θα λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά υπάρχουν πολλά σχέδια τα οποία θέλει να τονίσει. Γεωργία, λοιπόν, ε, ε, υπηρεσίες και ενέργεια. Συμφωνούμε λοιπόν για τη γεωργία, για τις βασικές παραμέτρους, για τη διαδικασία αυτή. Πώς ε, θα γίνει λοιπόν σωστή ανταλλαγή απόψεων. Θα πρέπει να υπάρχει προοδευτικότητα, συμμετρικότητα. Οι παράμετροι λοιπόν της διαπραγμάτευσης έχουν δημοσιευτεί Μιλούν για τη μεταβατική περίοδο, μιλούν για τα ευαίσθητα προϊόντα και τις σημαίες Αν εξετάσετε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία, θα υποβάλουμε και μία πρόσφορα η οποία είναι σημαντική και λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι στην Τινησία χρειάζεται πιο πολλές χρόνος για να γίνονται αυτές οι μεταρρυθμίσεις, αυτός ο εξυγχρονισμός. Επίσης, θα χορηγηθεί και βοήθεια προς την κατεύθυνση αυτή σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα και τις εξαγωγές. Αυτό θα ξεκινήσει φέτος με 90 εκατομμύρια ευρώ και αυτό θα επικεντρωθεί στους βασικούς τομείς του προγράμματος. Υποστήριξη λοιπόν χρηματοδοτική, στον τομέα τη ε, παροχή υπηρεσιών στη γεωργία και τεχνική αρρωγή αφετέρου. Θα είναι λοιπόν ευρύτερη η αρρωγή η οποία θα χορηγηθεί και οικονομική και τεχνική για τη γεωργία. Ένα τελευταίο στοιχείο. Αναφέρθηκε η σημασία της αλυσίδας αξίας και της αύξησης αυτής. Είχαμε λοιπόν κάποιους δείκτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε τι αφορά το ε, κεφάλαιο των γεωγραφικών ενδείξεων, είμαστε χαρούμενοι που πλέον ε, σα αναφέρουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη τη ΕΠΕΤΡΟΥ. Τώρα, να περάσω στο κεφάλαιο των υπηρεσιών. Για τον τομέα των υπηρεσιών, πράγματι έχουμε κάποιου κλάδου που είναι πολλά υποσχόμενοι από την ισιακή πλευρά και χαίρομαι για την έρευνα που έχει γίνει σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τι ψηφιακέ υπηρεσίε, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις τηλεπικοινωνίε. Εμεί από πλευρά μα οργανώνουμε και σχετικά εργαστήρια για το θέμα αυτό με την κοινωνία των πολιτών πριν τα τέλη του έτου, Αλλά αυτό που είναι επίση σαφέ είναι ότι σε ό,τι αφορά τι υπηρεσίε, η κινητικότητα των παρόχων υπηρεσιών για του οποίου θα ανοίξει η ευρωπαϊκή αγορά είναι πολύ σημαντική. Και γι' αυτό λοιπόν συνεργαζόμαστε στενά με του ε, συναδέλφου, σε ό,τι αφορά και τη Συμφωνία διευκόλυνση των Θεωρήσεων για να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν στενέ συνέργειε μεταξύ του DCFTA, του ΑΛΕΚΑ και τη διαδικασία διευκόλυνση θεωρήσεων. Τώρα, να στραφώ στην ενέργεια γιατί νομίζω ότι το ανέφερε και ο προηγούμενος ομιλητής. Στον τελευταίο γύρο η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε πρόταση για ένα φιλόδοξο κεφάλαιο για την ενέργεια και για πρώτες ανανεώσιμε ανανεώσιμες ενέργειες, μεγάλο κεφάλαιο και αυτό αναφέρεται και στην ιστοσελίδα μας. Ο στόχος είναι όχι μόνο να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει δίκαιο ανταγωνισμό, αλλά και να υποστηρίξουμε κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες έχει προεξαγγείλει την Ισία. Ξέρω ότι, ότι ο επικεφαλής της κυβέρνησης, ο κ. Σάιντ, επισκέφθηκε και τον Απρίλιο της Βρυξέλλας, παρουσίασε έναν οδικό χάρτη σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις σε προτεραιότητα. Και μία από τις κορυφαίες, λοιπόν, ε, ενέργειες από πλευρά της Τινησίας, που γραμματίζονται δηλαδή, είναι οι σχέδιο για την ενέργεια, που συνάδει με την Συμφωνία του Παρισιού. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίξει αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Γεωργικές, λοιπόν, υπηρεσίες, γεωργικά υπηρεσίες και ενέργεια. Τρεις τομείς ε, παραδειγματικοί. Και φυσικά τρίφεται και το θέμα του ενδιαφέροντος του από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντική αγορά τη Τινησία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε όμω εκεί για οικονομικού λόγου. Πιστεύουμε σε αυτή την εταιρική σχέση με του με τους ε, γείτονέ μα. Σήμερα δεν είναι ανοιχτή η γεωργική αγορά από αμφότερε τι πλευρέ. Άρα, προφανώς και ε, αντιπροσωπεύουμε τα συμφέροντα των εταιριών μας, των εξαγωγέων μας, ε, που πιστεύουν και ελπίζουν μέχρι το τέλο τη διαδικασία αυτή να μπορούν να εξαγάγουν με ευνοϊκού όρου. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Και θυμάμαι και τη συζήτηση για, τα, για τις ελιές και τα ελαιόδη προϊόντα. Θα δώσω το λόγο στην σκιώδη συγκητρία κυρία Λαλόντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Τζεριμπή και κύριε Νταούτ, ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, πληροφορίες που μας δώσατε, ε, για τις παρουσιάσεις σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα αυτά για τις διαπραγματεύσεις. Πολύ πρόσφατα γύρισα από την, την Ισία, πηγαίνω συχνά. Συμφωνώ με τα όσα είπε η κυρία Τζεριμπή για τα δικαιώματα των γυναικών, για την κοινωνία των πολιτών, όλες τις, ε, όλη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, αλλά και για τις απειλές ε, που επικρέμονται πάνω από τη χώρα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακούει πολύ προσεκτικά τα αιτήματα συμμετοχής των κοινωνία των πολιτών σε όλη τη διαδικασία, καθώς επίσης και της Βουλής της Τινησίας. Από την άλλη μεριά, το γεγονός ότι η η Γεωργία θα πρέπει να βγει ενισχυμένη από αυτή τη διαδικασία γιατί συνεισφέρει το 11% στο ΑΕΠ και 18% στις θέσεις εργασία. Επίσης ευχαριστώ την Κομισιόν που μας ενημέρωσε για τις εξελίξεις στο δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων. Ο τρίτος γύρος ε, προγραμματίζεται για το φθινόπωρο από ό,τι έχω καταλάβει ε, και ελπίζουμε ότι πριν το τέλος της θητείας μας θα υπάρχει μια πολιτική συμφωνία μεταξύ των διαπραγματευτών ω εισηγήτρια να ε, κάνω τι εξή παρατηρήσει. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά το πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε, δέκα χρόνια περίπου μετά την ε, Αραβική Άνοιξη, η Τινησία εδρεώνει την δημοκρατία της. Παρ' όλα αυτά, η, η όλη περιοχή χαρακτηρίζεται από αστάθεια, βρίσκεται πολύ κοντά στη Λιβύη και αυτό απειλεί την οικονομική ολοκλήρωση και δημιουργεί οικονομικά προβλήματα, είναι μεγάλο εμπόδιο στην ε, ορίμανση της δημοκρατίας. Η ανεργία των ε, νέων διπλωματούχων, για παράδειγμα, είναι τεράστια. 30% των νέων με δίπλωμα, με σημαντικό δίπλωμα, δεν έχουν δουλειά. Για το μέλλον της δημοκρατίας αυτό είναι πολύ απειλητικό. Θα πρέπει να ενδυναμώσουμε την οικονομία της ε, χώρας, να, να κάνουν πιο στενούς τους δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη μεριά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι την Ισία θα είναι μια ιστορία επιτυχίας για το Μαγκρέμπ έτσι ώστε και άλλες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμά της. Αυτό θα ευνοήσει την Τινησία αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να μην είναι ασύμετρη η ανάπτυξη. Θα πρέπει η κοινωνία των πολιτών να συμμετάσχει ισότιμα, το είπε ο κ. Νταβούτ δύο ερωτήσεις, μία στην Κομισιόν, αν έχω το χρόνο. Θα μπορούσε να μας διευκρινίσει τα της διάρθρωσης συμφωνίας για την κινητικότητα. Και μετά, στους δύο συμμετέχοντες, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές και πώς μπορούμε να επιτύχουμε σε αυτή τη συμφωνία στην εφαρμογή της. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσίκου. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Με πολύ μεγάλη προσοχή παρακολούθησα τις ε, δηλώσεις των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι προέβησαν σε μια εμβάθυνση, εις ανάλυση και φιλόδοξη όσο και θεμητή και σημαντική φιλοδοξία που εξέφρασαν με όλα αυτά τα στοιχεία που πρέπει να λάβει υπόψη η συμφωνία. Γεωργία, υπηρεσίες, κράτος δικαίου. Έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα πρόοδου η την Ισία τα τελευταία δέκα χρόνια και αυτά τα βήματα πρόοδου νομίζω τα οφείλει και στην ευαισθησία και την στήριξη που της προσέφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση χρόνια βέβαια τώρα υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε οικονομικούς όρους με στόχο τον εκδημοκρατισμό, την ε, πολιτική πρόοδο, την προαγωγή των πολιτικών δικαιωμάτων και νομίζω ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία που θα μας επέτρεπαν να ε, ελπίζουμε και για το μέλλον ακόμα καλύτερα πράγματα. Ταυτόχρονα ε, με ικανοποιούν και αυτά που είπε και η Επιτροπή, ότι δηλαδή έχουμε να κάνουμε όχι μόνο με μία προνομιούχο σχέση, δηλαδή την ε, αυστηρή τήρηση της συμφωνίας με όλα τα στοιχεία που έχει και την αμοιβαιότητα που προσφέρει χάρη στην ικανοποίηση στόχων και φιλοδοξιών που θέλουμε και εμείς ε, στην Ευρώπη αλλά και οι Τινήση να υλοποιήσουν. Ταυτόχρονα ε, αυτή η συμφωνία σημαίνει πρόοδο για την εκπαίδευση, για την γνώση, για την ψηφιακή οικονομία, την καινοτομία, την έρευνα. Έτσι λοιπόν προς τους εκπροσώπους και ιδιαίτερα τον εκπρόσωπο της ε, Γεωργίας, Έχουμε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Έχουμε ένα θέμα λεπτό και ευαίσθητο που είναι το θέμα του ελαιολάδου. Όταν έχουμε 70.000 τόνους σε ποσόστοση, από τις οποίες εσείς χρησιμοποιείτε 2.500 μόνο τόνους. Προφανώς απέχουμε, σε μεγάλο, ε, απέχουμε παρασάγκας από τις δυνατότητες που σας έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν βλέπω τι πρέπει να ε, καλύψει η συζήτηση για μια ενδεχόμενη παρέκκληση ή παράταση. Λοιπόν, ε, αυτές οι εξαιρετικές συνθήκες δεν μπορούν να, θεωρηθούν, να θεωρηθεί ότι ε, μονιμοποιούνται γιατί είναι εφάπαξ διευκολύνσεις. Ιδάλλως απλώς προχωρούμε σε μια μορφή υποστήριξης διαρκούς που δεν είναι υποφελής για κανέναν. Ο κύριος Μογέλ. Πρόεδρε ευχαριστώ. Η Αλεκά δεν είναι αυτός σκοπός. Η ομιλήτρια που ακούσαμε αυτό μας είπε. Είναι μια συμφωνία πάνω απ' όλα πολιτική έτσι τη βλέπουμε εμείς. Γιατί παρακολουθεί στην πορεία του μια χώρα στην πορεία της, μια χώρα που έδειξε υποδειγματική στάση κατά την δημοκρατική μετάβαση, που όμως αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά ε, σημαντικές οικονομικές αδυναμίες ή ευαισθησίες. Έτσι λοιπόν στηρίζουμε την, ε, την Ισία και βέβαια ε, ως εταίρο αλλά και μέσα από την πολιτική γειτονίας. Βεβαίω πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση πρώτα τη συμφωνία σύνδεση που προηγεί το της Αλέκα. Και για μένα τουλάχιστον ε, αυτό που λείπει είναι ότι δεν υπάρχει πραγματική ε, αξιολόγηση αντικτύπου της εφαρμογής της νέας αυτής συμφωνίας γιατί θα ήθελα να ξέρω εάν είναι σύμφωνη με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης που υποτιθώ ότι προάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά ακούμε να λέγεται ασυμμετρική και προοδευτική. Να εξασφαλιστεί πέστρος χρόνος μετάβασης. Μα είναι έτοιμη την Ισία. Έγινε λόγος για το τομέα της γεωργίας. Άκουσα τον ομιλητή από την ε, οργάνωση των γεωργών. Αλλά αν κοιτάξουμε την εικόνα που δίνει η γεωργία της ε, Τινησίας, ε, παρουσιάζει πολλά στοιχεία δυναμίας. Έτσι λοιπόν μια τέτοια συμφωνία καλό θα ήταν να μην ενισχύσει την αδυναμία ή το, την τροτότητα αυτού του τομέα. Αντίστοιχα με αυτά τα οποία βλέπουμε στην ΚΑΠ Φερρυπίν, στα, οπορι, ο, στα εσπεριδοειδή. Ήδη η Ισπανία, η οποία είναι από τις κύριες χώρες παραγωγής και εξαγωγής, έχει ακόμα σημαντική ε, σημαντικές δυσκολίες και, δεν έχει εγκαθιδρυθεί με τρόπο στεναρό ο τομέας της των εσπεριδοειδών. Μετά. Για την ρήτρα διατησίας βεβαίως πιστεύω ότι θα πρέπει να αποκλειστεί από τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ Τιτσιάνα. Ευχαριστώ κυρία Μπεγκίν. Η Τινησία είναι πολύ σημαντικός εταίρος για την Ευρώπη, κυρίως στη διάσταση της μετανάστευσης και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, επομένως με συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, που ήδη υφίσταται με την, ε, Τινησία βεβαίω βεβαίως και θα μπορούσε να βελτιωθεί, αλλά ταυτόχρονα συνεπάγεται και συμβασμούς που θα πρέπει με προσοχή να αξιολογήσουμε, κυρίως όσον αφορά την, ε, τον τομέα των γεωργικών για τα γεωργικά λοιπόν, πολύ σωστά όπως επεσήμανε και ο συνάδελφος, 10 χρόνια βλέπουμε ότι έχει πάνω από 50.000 τόνους ε, ποσόστος εξαγωγών για το λάδι ή την ωστόσο δεν, το έχει, δεν έχει αξιοποιήσει αυτές τις ε, ποσοστώσεις, αν και τον τελευταίο χρόνο έχει αυξηθεί ο όγκος των εξαγωγών της κατά 120%. Επομένως πρέπει να κοιτάξουμε και να αξιολογήσουμε μεγάλη προσοχή τι συνέπειες θα έχει μια τέτοια απόφαση για την ενίσχυση, διατήρηση των ε, εισαγωγών πολλό δε, από την Τινησία, πολλό δε μάλλον που δεν υπάρχει και καμία συμφωνία για τη σήμανση των προϊόντων ε, ελαίου στην Ευρώπη και θα μπορούσε και ο καταναλωτής αλλά και ο έμπορος να παραπλανηθεί. Ε, βεβαίως χαίρομαι πάντα όταν υπάρχει προστασία ικανοποιητική των ενδείξεων γεωγραφικής προελεύσεως ε, πρόκειται για μια συμφωνία φιλόδοξη οπωσδήποτε. Οι στόχοι ενδιαφέρουν όλες τις χώρες. Στόχος της προστασίας των εργαζομένων έχει τεράστια σημασία. Υπολείπεται αρκετά στην Τινησία και με όλα τα χαρακτηριστικά της οικονομίας, το ότι είναι εγγύς γεωγραφικά, το ότι έχει αδύναμο ε, νόμισμα, ε, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος εξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θέλω σε αυτό να μας καθησυχάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, και τώρα θα απαντήσουν ε, οι προσκεκλημένοι μας. Ο κύριος Ρίμπη πρώτα. Oui, merci beaucoup. Effectivement. Κυρία Ρίμπη, η αξιολόγηση των συμφωνιών ε, του 2014 των συμφωνιών σύνδεση εννοώ, ε, ήταν αντικείμενο συζήτησης και ε, με τις ε, οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών. Ε, γνωρίζετε, όπως είπαμε, ότι είμαστε σε μια κατάσταση σχετικής αστάθειας, χρειαζόμαστε χρόνο. Ο η διαχείριση του χρόνου είναι πολύ σημαντική. Πρόκειται για ε, συμφωνία η οποία θα επηρεάσει πολλές γενιές στο μέλλον. Γι' αυτό το λόγο προτιμάμε να ξεκινήσουμε με πιλωτικούς τομείς. Γιατί όχι. Όπως κάναμε με τις ε, υπηρεσίες ε, να αρχίσει να εφαρμόζεται το αυτό το κομμάτι της συμφωνίας, να αξιολογηθεί και να προχωρήσουμε σταδιακά. Είναι πιο ασφαλές. οι πολιτικοί στόχοι όπως ελέγχθη. οι ξένες ε, άμεσες επενδύσεις έχουν μειωθεί από το 2011. Λέω, το λέω προς τη συνάδελφό σας. Η κυρία Συγητρία λέει ότι επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση την Ισία να είναι η ιστορία επιτυχίας στο Μαγκρέμπ. Αυτό πρέπει να στηριχθεί με δράσεις, με πράξεις. Θα πρέπει να δοθεί κίνητρο για επενδύσεις στην Τινησία και να κινηθούμε προς ένα μοντέλο μεγαλύτερης τεχνολογικής μεταφοράς, μεταφοράς τεχνολογίας, συγγνώμη, περισσότερης καινοτομίας, απασχόλησης για τους διπλωματούχους και μια προσέγγιση η οποία θα ευνοεί την, την στον εκδημοκρατισμό της. Τι χρειάζεται, ρωτήθηκα συμμετοχική ε, συνεισφορά με τη συμμετοχή των επαγγελμάτων που έχουν άμεση σχέση με τις υπηρεσίες που εμπλέκονται άμεσα, που θα επηρεαστούν από την Συμφωνία ε, της Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες τους, να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους να βελτιωθεί η πρόσβασή τους στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τους πλαισιώσουμε. Και βέβαια η κινητικότητα. Το είπαμε και εξ αρχής αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Νταούτ. να απαντήσω στο, για το θέμα του ελαιολάδου. Το θέμα των ποσοστώσεων είναι κάτι το υποχρεωτικό. Οι ποσοστώσεις κατανέμονται στο χρόνο αλλά και, σε, και αναμήνα και αυτό είναι πολύ δύσκολο για μας. Επίση υπάρχουν πολύ μεγάλες αυξομοιώσεις ε, στην παραγωγή. Ε, είχαμε τρία χρόνια ξηρασίας που επηρέασε πάρα πολύ την παραγωγή μας κατά τη διάρκεια αυτών των ετών προφανώς δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε την χρήση όλων των ποσοστώσεών μας. Σε ό,τι αφορά το ότι μερικές φορές καταγγέλλονται νοθείες, να ξέρετε το εξής, η Τινησία εξαρτάται πάρα πολύ από το τι συμβαίνει στην Ισπανία, την Ιταλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες από πλευράς παραγωγής. Υπάρχει σημαντική παραγωγή ελαιολάδου στην Ευρώπη Οπότε αυτό μα δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην εξαγωγή του ελαιολάδου μα. Οπότε οι ποσοστό θα πρέπει να αναθεωρηθούν και όλο το καθεστώ θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Ε, η Τινησία θα κέρδιζε από την ε, ε, εδραίωση της ποιότητας ε, του ελαιολάδου, από την εδρώση της εικόνας καλής ποιότητας που θα πρέπει να έχει το ελαιολαδό μας. Έχουμε εξαιρετικά ε, ελαιόδεντρα, ανταλουσιανά, ε, 100 χρόνων και πάνω, πολλά από αυτά. Ε, οπότε έχουμε να κερδίσουμε από την πρόθεση της εικόνας ε, του ελαιολάδου και των ελιών. Οι ελιές μας είναι τελείως διαφορετικές από αυτές της Ευρώπης. Είναι σημαντικό λοιπόν να δουλέψουμε για αυτό το θέμα μαζί. Μελέτες επιπτώσεων πρέπει να γίνουν, να είναι σοβαρές και κοινέ. Θα πρέπει οι γνώσεις των δικών μας επιστημόνων να συνδυαστούν με αυτές των Ευρωπαίων. Ε, ένα έγγραφο για την Τινησία έκανε copy-paste ένα, από ένα έγγραφο του Μαρόκου ε, που αφορούσε το Μαρόκο για αυτό το θέμα. Δεν γίνεται αυτό. Θα πρέπει να... Οι μελέτες μας είναι ειδικά για την Τινησία. Τώρα, τι χρειάζεται. Πολιτική βούληση, διαφάνεια, συμπληρωματικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Μόνικα. Μάλιστα. Καταρχάς, να προσπαθήσω να απαντήσω στο ερώτημα της μελέτης δικτύπου γιατί υπήρξε μελέτη αντικτύπου για τη βιωσιμότητα πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Είναι δημόσιο το έγγραφο. Βέβαια, υπάρχουν σχέδια για μια πιο οριζόντια άσκηση στην Βουλή στην της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ε, εκτιμηθούν έξι από τα οκτώ FTAs και να ξεκινήσει η όλη διαδικασία, ελπίζουμε, στι αρχέ του επόμενου έτου. Στόχο μα θα ήταν να κοιτάξουμε όχι μόνο τι μεμονωμένε χώρε, εξπόστα έτσι, εκ των υστέρων, όχι εξάντα, αλλά για να διαπιστώσουμε ποιε είναι και οι βέλτιστε πρακτικέ, τα μαθήματα τα οποία διδαχθήκαμε από κάθε χώρα, γνωρίζοντα ότι είναι σε παρόμοιο επίπεδο πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά όλε οι χώρε. Για τι συνέργειε τώρα μεταξύ των δύο διαπραγματεύσεων. Είναι μοναδική ευκαιρία. Δεν είναι συχνά το, δεν παρουσιάζεται συχνά το φαινόμενο να έχουμε ε, διαπραγματεύσεις και για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων και για την ε, FTA και για την ε, εταιρική σχέση στον τομέα του Αυτό τι σημαίνει ότι θα έχουμε την κινητικότητα των ατόμων για να δίνουν τις υπηρεσίες. Χρειάζεται λοιπόν η παροχή υπηρεσιών, αλλά και να υπάρχει και αντίστοιχη θεώρηση για να μπορέσουν να μετακινηθούν. Αυτό που συμφωνήσαμε και συζητήσαμε στη συμφωνία για την διευκόλυνση των θεωρήσεων είναι η θεώρηση μέχρι 90 ημέρες στον χώρο Σέγγεν. Οτιδήποτε άλλο θα υπόκειται σε προτέρες συζητήσει. Αλλά θεωρούμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό από πλευρά ε, τη Τινησία, να υπάρχει ακριβώ αυτή η συνέργεια και γι' αυτό λοιπόν προγραμματίζουμε να προβούμε σε κοινέ συναντήσεις σε τα δύο κράτη με τα οποία γίνεται διαπραγμάτευση και τα κράτη-μέλη, προκειμένου να εξασφαλίσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Κάποιο ανέφερε το κεφάλαιο για την βιώσιμη ανάπτυξη του εμπορίου. Έπρεπε να το έχουμε φέρει το κεφάλαιο αυτό. Σημείωσε πολύ καλή πρόοδο και την ισιακή πλευρά. Φυσικά θέλει να αποδείξει ότι γίνονται σεβαστοί οι κανόνε για τη βιώσιμη ανάπτυξη και σε ό,τι αφορά και την Παγκόσμια Οργάνωση Εργασία. Το συγκριτικό πλεονέκτημα δεν είναι στην Τινησία το κόστος εργασία. Δεν μιλάμε για τον Μπαγκλαντέ ή άλλες τέτοιες χώρες. Όχι. Μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει στενό βαθμό, μεγάλο βαθμό ενσωμάτωσης με την ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας. Αυτά τα τρία ερωτήματα. Ευχαριστώ όλα και ο Πρόεδρος και έτσι ολοκληρώνεται το 13 της ημερήσιας διάταξης και είμαι βέβαιος ότι θα παρακολουθήσουμε με πολύ ενδιαφέρον και επισταμένος τις διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήλθατε από την Τινησία εδώ για να μας ενημερώσετε, να μας δώσετε τις πληροφορίες από πρώτο χέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και κάθε επιτυχία σας εύχομαι στις εργασίες. Το θέμα των υπηρεσιών τώρα. Υπηρεσίες Mode 5. Πώ να συμπεριλαμβάνετε δεσμεύσει για υπηρεσίε του τρόπου 5 στι διμερεί συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών και στο πολυμερέ στάδιο. Και δίνω το λόγο αμέσω στην Μαρίνα Πολτία να κάνει την παρουσίαση. Πέντε λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να... Αγαπητοί συνάδελφοι, ένα λεπτό λέει ο Πρόεδρος, ένα λεπτό. Σας παρακαλώ πολύ ησυχία, σας παρακαλώ πολύ ησυχία για να γίνει η παρουσίαση. Ο στόχος λοιπόν της μελέτης ήταν να εξετάσουμε το στόχο, τον τρόπο 5 της παροχής υπηρεσιών και κυρίως αυτών που προσφέρονται ε, από τομείς εκτός υπηρεσιών και σχετίζονται με διάφορα αγαθά επί παραδείγματι. Έχουν να κάνουν με το κατασκευαστικό κλάδο και τις υπηρεσίες που αναδεικνύονται τελευταία για να μιλήσουμε για τις χρηματοπιστωτικές μεταφορικές, επιμελητιακές, υπηρεσίες λογισμικού έρευνας ανάπτυξης περιβάλλοντος. Με ιδιαίτερη έμφαση στην servicification, την εισαγωγή της διάστασης της παροχής υπηρεσιών στην επιχειρηματική δραστηριότητα τόσο του πρωτογενούς όσο και του δευτερογενούς τομέα. Εδώ έχουμε να κάνουμε είτε με νέα στοιχεία που εισάγονται στην παραγωγή, την ε, σύνδεση υπηρεσιών ε, με, τα προϊόντα τους, την δεσμοποίηση προϊόντων και την ε, Ε, παροχή προϊόντων που είτε παράγονται μέσα στην επιχείρηση είτε έχουν ε, προκύψει από εξωτερική ανάθεση ε, είτε προκύπτουν σε υπεράκτιο επίπεδο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα λοιπόν. Ένα αυτοκίνητο. Όλοι ξέρουμε τι είναι το αυτοκίνητο. Εδώ βλέπετε τα τεχνικά του χαρακτηριστικά έχει διαφορούς ε, δέκτες ε, σε διάφορα σημεία, σχεδόν παντού γύρω-γύρω, για να βοηθήσει στην οδήγηση. Και με το παράδειγμα αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι η αξία του οχήματος αυτού απαρτίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες το περιεχόμενο των υπηρεσιών και το λογισμικό που τις προσφέρει. Εδώ είναι λοιπόν η αξία του προϊόντος. Και άρα τίθεται το ερώτημα εάν το προϊόν αυτό το χαρακτηρίζουμε ως αγαθό την ώρα που διασχίζει τα σύνορα ή όχι. Κάτι άλλο, ένα άλλο παράδειγμα, πιο παραδοσιακά προϊόντα Η ξυλία έχει κατά ποσοστό άνω του 50% περιεχόμενο υπηρεσίας που είναι η ξυλοκοπή, η μεταφορά, η ε, κοπή σε μικρότερα κομμάτια ή σε πριονίδι και το καθεξής. Άρα το ποσοστό της αξίας είναι πάρα πολύ μεγάλο στο αγαθό αυτό. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τη φρατζόλα. Για να παραχθεί μια φρατζόλα ψωμιού χρησιμοποιούνται αξίες, ε, υπηρεσίες, συγγνώμη, οποίες κατά την αξία τους ξεπερνούν το 72% του, της αξίας της φρατζόλας αυτής. Αν δούμε λοιπόν, ε, αν έρθει η ώρα να κάνουμε επιλογές ως προς την πολιτική, την εμπορική, θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η αξία της ε, υπηρεσίας σε αυτό τον κλάδο εμπορίου. Έχουμε μελέτες λοιπόν που μας δείχνουν ότι αυτός ο τρόπος 5 ε, αντιστοιχεί σε ποσοστό 20 έως και 47% μεριδίου αποδοτικότητας του τομέα και σε ένα σενάριο πολυμερές απελευθέρωσης των συναλλαγών, δηλαδή ένα σενάριο όπου τα προϊόντα αυτά δεν θα κατέβαλαν εισαγωγικού δασμούς, θα μιλούσαμε για ένα κέρδος ΑΕΠ, επί του ΑΕΠ έως το 2025 σε ύψος 300 δισεκατομμυρίων ευρώ ή όγκου εμπορίου αυξανόμενο κατά 500 δισεκατομμύρια ευρώ πάλι. Αρκετές χώρες θα μπορούσαν να κερδίσουν, βέβαια οι αναπτυσσόμενες περισσότερο, της Αφρικής, της Ασίας κτλ. Και βεβαίως η κλάδη της ε, παροχής υπηρεσιών σε βιομηχανικά ή άλλα κατεργασμένα προϊόντα θα απευθυνόνταν ιδιαίτερα. Θέσεις εργασίας. ...40% των ε, ε, προϊόντων που εξάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέονται με τον τρόπο 5. Αυτό όμως δεν ε, εξαντλείται εκεί γιατί έχουμε να κάνουμε και με πολλούς άλλους τρόπους διαμόρφωσης του προϊόντος, ε, πιο πράσινη οικονομία, τη στρατηγική του 2020 ουσιαστικά, πιο ευφυή οικονομία, περιβαλλοντικά προϊόντα και υπηρεσίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις συμμετέχουν εξαγωγικό δυναμικό, παραγωγικότητα συνολική. Ποιες είναι οι προκλήσεις λοιπόν που μας φέρνει αυτός ο τρόπος 5. Επαναλαμβάνω ότι δεν πρόκειται για αναγνωρισμένο υπό την GATS ε, τρόπο παροχής μιας υπηρεσίας. Δεν είναι αναγνωρισμένος επαναλαμβάνω και ως εκ τούτου συναλλαγές, εισαγωγές ή εξαγωγικές που καταγράφουμε υφίστανται τους ε, εισαγωγικούς δασμούς ή τις ποσοστώσεις που προβλέπονται για τα προϊόντα, τα υλικά προϊόντα. Και αυτό έχει να κάνει και με το, αυτό το βλέπουμε να αντικατοπτρίστε και στους κανόνες για την προέλευση των ε, συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών. με δυσμενή προφανώς, δυσμενείς συνέπειες για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές και τις υπηρεσίες τρόπου 5. Κυρία, ευρήματα. Προσοχή πρέπει να δώσουμε πάνω απ' όλα στην απελευθέρωση αυτών των προϊόντων ε, για να καλυφθούν τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, εκεί πρέπει να δώσουμε την έμφαση στις υπηρεσίες τρόπο 5. Επίσης ε, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, δεν θα έπρεπε να αποκλείσουμε μία ε, δυνατότητα για γενικές πολυμερείς διαπραγματεύσεις που θα απελευθέρωναν και αυτές τις συνολικές αλυσίδες αξίας όπως τις ονομάζουμε, GVC, σε παιδοποέ. Ε, μια προκαταρκτική ε, περιγραφή, ένας προκαταρκτικός ορισμός πάνω απ' όλα είναι απαραίτητος και μια και δεν υπάρχει. Εμείς θα προτείναμε ότι αυτές οι υπηρεσίες τρόπου 5 είναι υπηρεσίες που συμπληρώνονται ή συνδέονται με αγαθά των οποίων η αξία και η προέλευση μπορεί να ε, ανοιχνευθεί από την αξιολόγηση στο τελωνίο των αντίστοιχων αγαθών ε, επιλογές ο Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, διμερής ή πολυμερής, τι μπορεί να γίνει δηλαδή σε επίπεδο ΠΟΕ, τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο δίμερες, ε, Συμφωνίων Ελεύθερων Συναλλαγών. Έχουμε λοιπόν αναζητήσει και βρει τις εξής επιλογές που είναι καταρχάς έκπτωση δασμού σε επίπεδο τελωνίων ε, με βάση και τη συμφωνία αξιολόγησης ή τιμολόγησης ε, που επιτρέπει την ε, απαλλαγή μέρους της αξίας από την τελωνιακή δήλωση που έχει σαν συνέπεια την ε, καταβολή πιο μικρών τελωνιακών δασμών. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει προβλεφθεί αυτό για την απελευθέρωση των υπηρεσιών. Μετά έχουμε μια άλλη εξαίρεση που προβλέπεται για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ίσως μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευση. Ωστόσο εδώ δεν ε, υπάγεται στην παγκόσμια οργάνωση των τελωνίων Πάντως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως έμπνευση και μετά μια γενική συνθήκη, των ε, σύμβαση των, ε, της αλυσίδας αξίας, GVC δηλαδή, που θα μπορούσαμε να ε, διεκδικήσουμε, να επιδιώξουμε σε πεδοπολιμερές Ε, τελωνιακή δεσμία και μείωσή τους, εάν σε πεδοποέ δεν εξασφαλιστεί, μπορούμε να την επιδιώξουμε σε πεδοδημερών συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών θα ήταν πιο εύκολο κάτι τέτοιο και θα μπορούσαμε και συμπληρωματικά να, να συμπεριλάβουμε έναν ε, όρο γεωγραφικής προελεύσεως που θα μπορούσε να ήταν ε, σαφής και ε, χρήσιμος. Και τελικά ε, συστάσεις, πρώτα πρέπει να περιγράψουμε αυτές τις υπηρεσίες τρόπο 5, να αντιληφθούμε τι συνέπειες έχουν και τι χαρακτηριστικά, να αναπτύξουμε συμπληρωματικές οικονομικές αναλύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον κόσμο, να θεσπίσουμε μια ομάδα έργα εμπειρογνωμόνων ε, υπηρεσιών τρίπου, τρόπου 5, να ευαισθητοποιήσουμε τον ιδιωτικό τομέα στις χώρες μέλη, μέλη που ενδεχομένως δεν ήθελαν να υποστηρίξουν, συνεργασία με διάφορους οργανισμούς διεθνείς που έχουν ήδη ξεκινήσει σχετική δουλειά και μια χαρτογράφηση των ε, δεδομένων και δυνατών επιλογών. Ως προς την έρευνα στο μέλλον, βεβαίως η έκθεσή μας είναι μια πρώτη ε, προσπάθεια. Βεβαίως ε, χρειαζόμαστε πιο ουσιαστικές μελέτες, ε, όχι μόνο το παράδειγμα που σας έδωσα με τη φρατζόλα και το αυτοκίνητο ή το iPhone. Χρειάζεται οπωσδήποτε περισσότερη μελέτη και ανάλυση, ιδιαίτερα για χώρες αναπτυσσόμενες που μπορεί να μην δείξουν ιδιαίτερη διάθεση να υιοθετήσουν την ιδέα αμέσως. Πάντως θα πρέπει να επιδιωχθεί σε πολυμερές επίπεδο ΠΟΕ ή και εκτός ΠΟΕ ε, μια σύμβαση, μια συμφωνία για την αλυσίδα αξιών, εάν στο επίπεδο του ΠΟΕ είναι πρόβλημα το σύστημα λήψης αποφάσεων οπωσδήποτε εκτός αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρονται όλα αυτά για τι ψηφιακέ εξελίξεις Το αυτόνομο αυτοκίνητο θα πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο αργότερα. Δύο λεπτά στην Κομισιόν. Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε πρώτα, γιατί πολλοί συνάδελφοι ήρθαν για να ψηφίσουν. Θα μας πάρει μισή ώρα. Όχι, όχι, έχουμε την ημερήσια διαταξή μας. Αν, αν όλοι ήταν εδώ στις 9 δεν θα είχαμε πρόβλημα, θα είχαμε ήδη τελειώσει. Λοιπόν, να θυμάστε τις παρουσίες εσείς εγκαίρως. Παρακαλώ, Κομισιόν. Ε, καλωσορίζω την ε, πρωτοβουλία σας για να συζητήσετε επισήμως ε, το θέμα του τρόπου 5 ε, και είναι σημαντική αυτή η συζήτηση, αυτός ο τρόπος, τρόπος 5, είναι πολύ σημαντικός διότι έχει άμεση σχέση με την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Είτε το αντιλαμβανόμαστε πλήρως είτε όχι. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον, την συγγήτρια της έκθεσης. Έχουμε πολλές εναλλακτικές μπροστά μας, άλλες είναι πιο φιλόδοξες, λιγότερο. Πάντως ε, είναι πολλά υποσχόμενες ε, σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα επί των οικονομικών παραγόντων μας και των οικονομικών φορέων μας. Ε, πάρα πολλοί εξαγωγείς μας ενδιαφέρονται να σημειώσουμε πρόοδο σε ό,τι αφορά τον τρόπο 5. Όχι μόνο παρόχοι υπηρεσιών, αλλά και πολλοί βιομηχανικοί παίκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξαρτώνται από την εξωτερική ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα του, των υπηρεσιών του τρόπου 5. Είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κλειδί και η κατάσταση σίγουρα δεν είναι βέλτιστη. Θέλω να υπογραμμίσω δύο πράγματα που εξηγούνται στην έκθεση, αλλά καλό είναι να τα υπογραμμίσουμε. Πρώτον, δείχνει να είναι μια καινούρια έννοια, αλλά διατάξεις για τον τρόπο 5 ε, δεν είναι κάτι καινούριο εφαρμόζονται οι αντίστοιχε διατάξεις από τους ελληνικού μας υπαλλήλους τα τελευταία 30 χρόνια στις αγωγέ. Οπότε υφίστανται δρεωμένε διαδικασίες. Οι Ευρωπαίοι τελωνιακοί υπάλληλοι έχουν την δυνατότητα να απομειώσουν την ε, τελωνιακή αξία των υπηρεσιών αυτών αν πληρούνται τα κριτήρια του αντίστοιχου άρθρου. Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι να ε, επεκταθεί η εφαρμογή του και στις εξαγωγές. Παρόλο ότι σε πολυμερές επίπεδο είναι δύσκολο να προωθεί αυτή η ιδέα, γιατί θα ευνοούσε μεν όλο τον κόσμο, αλλά θα έπρεπε πρώτα να αποδειχθεί η αξία της ιδέας σε μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών και μετά να επεκταθεί σε όλο τον κόσμο. Άλλες παρατηρήσεις? Κύριε Μινέ. Να πω κι εγώ δύο λόγια. Επιτρέπετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ να εκφράσω την εναλλαγή μου με τους διερμηνείς οι οποίοι συνεχίζουν την κινητοποίησή τους. Πρόεδρε, το κόμμα μου ανησυχεί για την ε, παγκόσμια απελευθέρωση των υπηρεσιών. Ε, χρησιμοποιούνται ουσιαστικά οι εργαζόμενοι και συγκριτικό πλεονέκτημα τι σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνεται κάθε συναλλαγή με τον πιο ε, α, τρόπο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι πιο ελκυστικοί είναι οι εργαζόμενοι που πληρώνονται χαμηλότερα, όπου υπάρχουν ε, τα χαμηλότερο κόστος για καλές ε, όμως ε, συνθήκες εργασίας. Αυτό ίσως να είναι καλό για τον καταναλωτή και για τον εργοδότη, όχι όμως για τον εργαζόμενο. δεν έχει σημασία μόνο πόσα μπορούμε να αγοράσουμε με τα χρήματά μας. ότι αφορά λοιπόν την απελευθέρωση των ε, συμφωνιών και έτσι καταλαβαίνω τι γίνεται, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς ποιε είναι οι συνέπειες. Τι ερωτήσει έχω να κάνω. Καταρχά. θα γίνει μελέτη αντικτύπου για να εξεταστούν ε, οι συνέπειε των προτάσεων. Και δεύτερη ερώτηση σε ό,τι αφορά το crime working την παροχή δηλαδή υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως κάνει η Amazon για παράδειγμα. Υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ Mode 5, τρόπου 5 και crowd working. Υπάρχει περαιτέρω απελευθέρωση. Αυτό θα είναι κακή είδηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Άλλα σχόλια όχι. Μάλιστα. Και κλείνει δυστυχώ το μικρόφωνο του Πρόεδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας και τα σχόλιά σας. Σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας και τη μελέτη δικτύπου, όπως έλεγα και στην παρουσίαση, αυτή η έκθεση αποτελεί μόνο μία πρώτη φάση. Η μελέτη και οι συζητήσεις είναι ακόμα σε πρώιμη φάση. Και ένα από τα ευρήματα ήταν η δημιουργία μιας ομάδας εμπεριαγνωμόνων που θα χαρτογραφήσουν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να είναι υπό ανάλυση και η μελέτη αντικτύπου υλοποιήσω. Λοιπόν, ε, φαντάζομαι ότι θα είναι ένα θέμα για το crowd working και τη σχέση του με τον τρόπο 5, mode 5. Δεν ήταν αυτό ακόμα τμήμα της ε, συζήτησης. Αν υπάρξει όμως ομάδα, προφανώς θα δώσει εντολή για την ενέργεια άλλων α, ε, ε, ερευνών για να έχουμε πιο πολλά στοιχεία για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και προφανώς θα συνεχίσουμε τις συζήτηση για το Mold 5. και όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία θα μα απασχολήσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και έτσι ολοκληρώνεται το σημείο 14 στην ημερησία διάταξη. Και πρωτού περάσουμε στο σημείο 15 και τις ε, ψηφοφορίε, να πω χρόνια πολλά στα Χλίμου Τσόλτ. Έχετε γενέθλιά του. Χρόνια πολλά. 38, I guess. So. Τα 38 φαντάζομαι κλείνεται. 15 will be the... Στο 15. Πρώτη ψηφοφορία. Να κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση πριν το ξεκινήσουμε. Παρακαλώ ψηφίζουμε δοκιμαστικά. Everybody voted. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. παρακαλώ τη ψηφοφορία. Μάλιστα. Όλα εντάξει, να ξεκινήσουμε στο σημείο 15 λοιπόν τη ημερησία διαταξή. Μία ψηφοφορία μόνο. Έναξη ψηφοφορία. Πέρασε. εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. συγκαρτηρία στον κύριο Κασπάρη. Στο σημείο 16 έχουμε προφορική ερώτηση με την ΔΕΒΕ ε, και αυτό μία και μοναδική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Και πέρασε. Εγκρίθηκε. Μεγάλη πλειοψηφία στο 17 ψήφισμα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μολδαβία. Τροπολογία 3. Σε δύο τμήματα, παρακαλώ. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Τροπολογία. Αποχές ε, απορρίπτεται. Τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε 5 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε η 6 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε 7 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε 7 8 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε 9 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε η 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Προφορική τροπολογία της κυρίας Χάουταλα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. πίπτη η 11. 12 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Η ένα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορριφθήκε. Δύο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκριθήκε. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Παρακαλώ ψηφίζουμε. Και πέρασε. ευρια η πλειοψηφία υπέρ εγκρίθηκε συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και τώρα στο σημείο 18 έχουμε και πάλι ψήφιση για την εφαρμογή της Συμφωνίας τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Γεωργία αυτή τη φορά. Η τροπολογία 1 υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίθηκε. 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 5 υπέρ κατά άποχες έλεγχος να ελέγξουμε παρακαλώ την τροπολογία 9, 5 συγγνώμη ψηφίζουμε και πέρα της τροπολογίας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε η 6 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβαστική. 1 ειπε κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 15 ειπε κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές Εγκρίθηκε. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 21 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίθηκε. 23 υπέρ. Κατά.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 αποχές εγκρίθηκε και τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ έναρξη ψηφοφορίας και πέρασε και αυτή εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία συγχαρητήρια στο 19 και πάλι ψήφισμα με την συμφωνία σύνδεση αυτή τη φορά με την Ουκρανία και η τροπολογία 1 είναι η πρώτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά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 Περνάμε τώρα στο σημείο 20. Κατάσταση των σχέσεων Ευρωπαϊκή Ένωση και ΙΠΑ. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 27 28, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 28 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. και 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. πίπτη 39 λοιπόν υπέρ κατά άποχες. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά κάνουμε παρακαλώ έναν ηλεκτρονικό έλεγχο. Δεν είναι απόλυτα σαφές. Ψηφίζουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Για την 39. Πέρας. Α, εγκρίνεται με σαφήνεια. Σας παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας. 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. και 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται συμβαστική 8α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ψηφίζουμε παρακαλώ την 67 Απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας ελέγξουμε και την 68, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Και ψηφίζουμε το ψήφισμα στο σύνολό του ηλεκτρονικά αυτή τη φορά. Ψηφίζουμε. Πέρας. Και αυτό εγκρίθηκε με ευρία ψηφοφορία. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ε, and Ευχαριστώ για την πολύ καλή συνεργασία, λέει η συγγήτρια. 21. Σημείο 21 της ημέρης της διάταξης. Ε, προστήκη στο ψήφισμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφγανιστάν. Ενιά ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Ε, ωραία, υπερψηφίστηκε. Περνάμε στο σημείο 22. Παρακολούθηση δραστηριοτήτων ομάδων. Σημαντικό τμήμα των εργασιών μας. Όποιος θέλει να φύγει παρακαλώ πολύ ήσυχα ήσυχα ακροποδητή. Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των ομάδων μας είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Καταρχήν ξεκινούμε με την Νότια Αφρική. Άντια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Παρακολουθεί. Έχουμε μια συμφωνία με την Κοινότητα ανάπτυξη νότια Αφρική. Συναντηθήκαμε η παρουσία του Γενική Διεύθυνση Trade και των εκπροσώπων τη ΟΚΕ. Η Κομισιόν μα ενημέρωσε για την εφαρμογή τη συμφωνία που υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2016 και άρχισε να εφαρμόζεται προσωρινά τον Οκτώβριο του 2016. Είναι εμπορική συμφωνία με τις χώρες Μποτσουάνα, Λεζότο, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Νότια Αφρική και Σουαζιλάνδη. Η Νότια Αφρική προφανώ είναι ο πιο ισχυρό εταίρο στην περιοχή. Είναι χώρε που αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικέ προκλήσει. Η Μοζαμβίκη και το Λεσότο είναι από τι λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε. Η εφαρμογή τη συμφωνία ε, έχει αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα συντονισμού ε, στο εσωτερικό της, της περιοχής, στον χώρο της περιοχής. Βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη, η απουσία κοινή πλατφόρμας τη κοινωνία των πολιτών σε αυτές τις χώρες. ο διάλογος με, τις κοινωνίες, με την κοινωνία των πολιτών, μεταξύ κοινωνίας πολιτών και κυβερνήσεων σε πολλές από αυτές τις χώρες είναι πολύ αδυνάμος. Επίσης, δυστυχώς έχουμε σημαντικά, κάποια σημαντικά εμπορικά προβλήματα τα οποία κρεμούν. Η, η, ε, η Τελωνιακή Ένωση της Νότιας Αφρικής, ε, των χώρων της Νότιας Αφρικής, συγγνώμη, τις Νότιας Αφρικής χώρα ε, αύξησε του δασμούς σε 600 γεωργικά προβλήματα, ε, σε 600 ε, προϊόντα εφαντουργικά. το κοινή υπουργική συνάντηση θα λάβει χώρα το Φεβρουάριο του 2019. Τι θα είναι η επόμενη εξέλιξη. Παρακαλώ πολύ, ερωτήσεις, παρατηρήσεις. Όχι. Στις 5 Ιουνίου έλαβε χώρα η συνάντηση ομάδα παρακολούθησης συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Νομίζω όμως ότι συζητήθηκαν τα ίδια θέματα που συζητήσαμε χτες με τον κύριο Ντεμαρτή. και η εξοεδαφική επίπτωση που επίσης συζητήσαμε με την κυρία Νίντια χτες. Οπότε εκεί δεν έχουμε άλλες πληροφορίες να δώσουμε. Ε, ομάδα παρακολούθησης με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής. Την τρίτη συνήλθε η ομάδα παρακολούθησης. Παρουσία του Πρόεδρου κ. Του, παρουσία του κ. Γιώργενσεν από την Κομισιόν του πρέσβη Φάρο από την Κωνσταντίνα που ε, προεδρεύει τη ΣΥΚΑ. Καταρχήν, ένα πρόβλημα που έχουμε αντιμετωπίσει επανειλημμένο στο παρελθόν. Γνωρίζετε ότι το 2019 θα γίνει η αξιολόγηση του λειτουργία ιδιαίτερα του εμπορικού πυλώνα. Η Συμφωνία Σύνδεση υπάρχει εδώ και πέντε χρόνια, λειτουργεί εδώ και πέντε χρόνια ε, σε ό,τι αφορά την προσωρινή εφαρμογή του εμπορικού πυλώνα, αλλά μέχρι τώρα τέσσερα κράτη-μέλη δεν την έχουν επικυρώσει. Θυμάμαι ότι και εσείς και κάποιοι άλλοι πρόεδροι γράψατε μια επιστολή στον πρόεδρο Ταγιάννη για να του επιστήσετε την προσοχή στο θέμα αυτό προκειμένου ε, βουλευτές από διάφορα κράτη, ε, συγγνώμη, τα, προκειμένου να πιεστούν τα κοινοβούλια αυτών των κρατών μελών να επιταχύνουν. Υπάρχουν ε, βέβαια πολύ περίπλοκα θέματα που πρέπει να εξεταστούν σε βάθος, όμως να παίρνει και παραπάνω πέντε χρόνια για να επικυρωθεί μια συμφωνία. Πώς μπορούμε να χτίσουμε εμπιστοσύνη σε ένα γρήγορα μεταβαλλόμενο κόσμο με αυτόν τον τρόπο. Οπότε θα πρέπει να βρούμε ένα καλύτερο μηχανισμό συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Εδώ τω μεταξύ, έλαμε χώρα τέσσερις συναντήσεις ε, του ε, και άλλων επιτροπών. Την περασμένη εβδομάδα μία από τις αυτές επιτροπές ε, συναντήθηκε έχουμε κάποιες θετικές και κάποιες, κάποια θετικά σημεία και κάποια αρνητικά. Η Κομισιόν μας ε, παρουσίασε τις αξιολογήσεις της μέσω εκθέσεων. Οι εμπορικές ροές εξέλισσονται ικανοποιητικά. Η αύξηση είναι μικρή, αλλά όχι όμως όσο άλλες ροές παρόμοιες. Αν δούμε τις εξαγωγές από τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής, μπανάνα, φινικέλαιο, ψάρια, καφές, αρκετά δυναμικά, ιδιαίτερα η Κώστα Ρίκα, ε, ιατρικό εξοπλισμό και φινικέλαιο κυρίως, εστιάζονται όμως σε συγκεκριμένους κλάδους. Και οι, οι τελωνικέ ε, ποσοστό χωρί δασμού δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πλήρω Καθ' ολοκλήρια. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούν μόνο ε, το, ε, το 100% μόνο στο, ε, στη ζάχαρη και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί 50 ή 75% σε, για στο αποκορυφωμένο γάλα, σε σκόνη, το γάλα κλπ. Οπότε δεν τις, ούτε εμεί χρησιμοποιούμε πλήρως τις ποσοστώσεις μας θα ήταν πολύ σημαντικό να δούμε ποιοι είναι οι λόγοι πίσω από αυτό. Υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης, υπάρχει ένα θέμα τιμών, υπάρχουν εσωτερικά προβλήματα που παρεμποδίζουν τις εξαγωγές. Πρέπει να το συζητήσουμε. Έχουμε βέβαια και εμπόδια, για παράδειγμα φορολογία στην Κωνσταντίνα, ε, τέλεια τη χρήση σκάνερ στην Ικαράγουα, ε, δίκαιο του ανταγωνισμού που δεν έχει πλήρως ε, εξυγχρονιστεί σε άλλες χώρες. Έχουμε δομέ διαλόγου με κάποιες από τις χώρες αυτές, με την κοινωνία των πολιτών, αλλά όχι με όλες. Η Κομισιόν είπε ότι παρακολουθεί κάθε μία από αυτέ τι περιπτώσει χωριστά με κάθε χώρα. Για παράδειγμα έχουν ξεκινήσει με τη Γουατεμάλα. συνάδελφοι κατά τη διάρκεια τη συζήτηση με τον πρέσβη ανέφεραν ότι υπάρχουν μεγάλε διαφορέ ανάμεσα σε χώρε, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών. Μικρομεσαίε επιχειρήσει δεν αναφέρονται ρητά στη συμφωνία και αυτό είναι ένα πρόβλημα, θα πρέπει να το συζητήσουμε. Η Κομισιόν σημείωσε την ανάγκη να προχωρήσει η περιφερειακή ολοκλήρωση. Όλα αυτά πολύ καλά βέβαια. Ε, οι επικρίσεις είναι εύκολες, αλλά αν δούμε τι σημαίνει και στο εσωτερικό της ευρωπαϊκή Ένωσης, όσο θα έπρεπε να είμαστε πιο ταπεινοί. ορισμένες ιδέες για την έκθεση πρωτοβουλίας είναι η Ε, μάλλον θα τις έχουμε μετά τις ε, ε, διακοπές, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για διαφοροποίηση της οικονομίας, για ποιους λόγους ε, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πλήρω οι ποσοστό και ευκαιρίε που δίνονται, το θέμα τη ε, επικύρωσης, επικύρωση, μείωση των φραγμών στο εμπόριο και ε, βελτίωση τη δουλειά μα σε ό,τι αφορά τα εργασιακά δικαιώματα και προώθηση τη περιφερειακή ολοκλήρωση. Αυτά είναι τα βασικά σημεία τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην έκθεση πρωτοβουλία. Θα περιμένουμε να δούμε το κείμενο μετά το καλοκαίρι και να σχολιάσουμε. Ευχαριστώ πολύ για την ε, πληρέστατη αυτή επισκόπηση. Οι παρατηρήσεις, οι ερωτήσεις παρακαλώ. Άρα, να προχωρήσουμε σε περισσότερες δράσεις για την ε, κύρωση, να διευκολύνουμε τα κράτη-μέρη να πάρουν τη σχετική απόφαση. Οι λοιπές χώρες, 19 Ιουνίου και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, είχαμε χτες μια διεξοδική συζήτηση για διάφορες πτυχές των λατινοαμερικανικών χωρών και έτσι θα προσπαθήσω να είμαστε εδώ πιο σύντομος και ο εισηγητής ε, για, για τη Συμφωνία Περού και Κολομβίας παρουσίασε χτες μόλις τις ιδέες του για, τα, για, την έκθεση, για την έκθεση εφαρμογής ε, κατά τα πρώτα πέντε χρόνια της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Περού Κολομβίας. Σε δύο τμήματα για, την, για το Περού και την Κολομβία την πρώτη πενταετία και τον ένα χρόνο της πρόσβασης του Εκουαδόρ. Μιλήσαμε και με τον κύριο Γιώργενσεν. Ε, ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε στο ζήτημα του συστήματος συνοικευμένων προτιμήσεων και τις εξελίξεις σε σχέση με το Περού και την Κολομβία φέτος Κάποιες ε, πτυχές ε, του κεφαλαίου TST παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με την υλοποίηση. Επομένως, ε, πραγματοποίηση του οδικού χάρτη στο Εκουαδόρ. Βλέπουμε την βούληση της χώρας να επιταχύνει μια συμφωνία ειδική και άλλωστε να αντικατοπτρίζει και τις διμερείς, ε, πολλές διμερείς που είχε στο παρελθόν με χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Εκουαδόρ, επιμέρους συμφωνίας. Τώρα θέλει συνολική και επίσης θα ήταν ίσως πιο σημαντικό για τα βιολογικά προϊόντα ε, αντίστοιχη με αυτή που έχουμε και με τη Χιλή ε, για την ενίσχυση λοιπόν των συναλλαγών στο βιολογικό ε, στο βιολογικό κλάδο όπου είναι και πολύ ανταγωνιστικό σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση το Εκουαδόρ στην οργάνωση των μελλοντικών ε, εμπορικών συναλλαγών. Θα έχει σημασία αυτό. Ίσως και κάποιες πτυχές εμπορικών σχέσεων που δεν έχουν να κάνουν με, την, με τις παραδοσιακές μορφές ανάπτυξης και εμπορίου. Αλλά θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη δυνατότητα της αύξησης του μεριδίου αγοράς σε βιολογικά προϊόντα των χωρών αυτών έτσι ώστε να μπορέσουν να ανοίξουν περισσότερο το χώρο που καταλαμβάνουν στη διεθνή αγορά. Επίσης συναντηθήκαμε με εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων παραγωγών μπανάνας του Εκουαδόρ αλλά και αντίστοιχα εκπροσώπων συνδικάτων ε, του κλάδου μπανάνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταγράφουν ε, μία μη ικανοποιητική κατάσταση σε αρκετούς τομείς στην ε, παραγωγή μπανάνας. Και είπαμε πώς θα μπορούσαμε να δώσουμε μια απάντηση υπεύθυνη και την υποστήριξη μιας οργανωμένης ε, παραγωγής για τις μεγαλύτερες ε, επιχειρήσεις, αλλά ταυτόχρονα και να ε, συμβάλλουμε στη συνεργασία με τις κυβερνήσεις αφενός, αλλά και τις συμβουλευτικές ομάδες αφετέρου, δηλαδή να στηρίξουμε τις κυβερνήσεις στην προσπάθεια να συνεχίσουν τον αγώνα. και σε οικολογικό επίπεδο για την υλοποίηση αυτού του, κομμάτου, του, του κομματιού του τμήματος της συμφωνίας. Η ομάδα λοιπόν συμβουλών θα παρακολουθεί στην περαιτέρω ε, η ε, τήρηση των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών και την υλοποίησή τους, ε, υλοποίησή της, δεν χρειάζεται να περιμένουμε άλλα πέντε χρόνια βέβαια για το Εκουαδόρ. Αντιθέτω, θα έπρεπε να επιταχύνουμε στο δυνατόν αυτή τη φάση, την πρώτη φάση εισαγωγή ε, και υλοποίηση και να παρακολουθούμε πώ εξελίσσεται. Παρακαλώ, ερωτήσει ή παρατηρήσει. Ναι, ευχαριστώ και πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ για την ε, έκθεση αυτή. Αυτά που είπατε για την παραγωγή μπανάνας ε, στο Εκουαδόρ με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα γιατί βλέπουμε από το Ηνωμένο Βασίλειο άρθρα σχετικά με το ε, με τις συνέπειες στον ε, ευρωπαϊκό κλάδο μπανάνας, μάλλον τον ε, βρετανικό κλάδο μπανάνας. Καλό θα ήταν λοιπόν να παρακολουθήσουμε τι κάνουν οι συμβουλευτικές αυτές ομάδες και αν συζητούν το συγκεκριμένο θέμα ή όχι. Θες να απαντήσεις? Ναι, συμφωνώ απολύτως με την παρατήρηση του David γιατί πρέπει πιστεύω να είναι και η δουλειά αυτή κυρίως της συμβουλευτικής ομάδας καθώς υπάρχουν πολλές εξελίξεις. Μπορεί στο Περού να μην έχουμε ακόμα εγκαθιδρύσει μια τέτοια συμβουλευτική ομάδα. Ένα από τα μαθήματα που αποκομίσαμε με την επίσκεψή μας εκεί. Η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Επιτροπής ε, και η λοιποί τη συμβουλευτική ομάδα από ευρωπαϊκή πλευρά επιμένουν πριν πάει στο Συμβούλιο που σχεδιάζεται για τον Νοέμβριο του 2018 στο Κίτο για τις τρεις χώρες να έχει προηγηθεί συνεδρίαση και κοινή ίσως των συμβουλευτικών ομάδων ώστε να τεθούν επιτάπητος όλα τα ζητήματα και να δούμε πόσο απέχουμε ή πόσο μπορούμε να πλησιάσουμε. Γιατί είναι μερικές φορές οι πληροφορίες από τα Υπουργεία αντιφατικές. Δηλαδή άλλη εικόνα μας δίνουν τα συνδικάτα, άλλα οι κυβερνήσεις, ε, οι οργανώσεις των πολιτών, άλλα οι εκπρόσωποι των ε, ε και ούτω καθεξής. Άρα χρειάζεται μια συνεργασία, συνεννόηση, ευθύνη. Αυτό το είπαμε και στην ομάδα παρακολούθησης την Τρίτη. Ακολουθούμε τον κύριο Φύσης εδώ και τους δύο εισηγητές δηλαδή στην πρόταση να παρακολουθήσουμε τι συμβαίνει, να προσπαθήσουμε να διαρευνήσουμε τι συμβαίνει, να ρωτήσουμε και την Επιτροπή για το τι θα γίνει ε, σε σχέση με συνεδριάσεις των Συμβουλευτικών Επιτροπών μέχρι τον Νοέμβριο. Καλώς λέει ο πρόεδρο. αν δεν ζητεί κανεί άλλο το λόγο, στο λόγο κλείνουμε και το σημείο 22 και πάμε στο σημείο 23. Η αντίδρασή μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την τη θάσευση της παγκοσμιοποίηση σε πτυχές. Η κυρία Μόσκα. Ναι, αντικαθιστώ τον Γιάκεμ Σούστερ, ο οποίο είναι συγκεκριτής μα. Να διαβάσω τα σχόλιά του. Αγαπητοί συνάδελφοι, αντιμετωπίζουμε ακόμα θέματα αντιπαγκοσμιοποίησης και τα θέματα αυτά είναι πάρα πολύ σύνθετα. Έχουν αναδιαρθρώσει την ε, κατανομή της κατανομή ε, εργασίας καθώς και την ανεξάρτηση των χωρών. Τα ωφέλη δεν κατανέμονται ισότιμα μεταξύ περιφερειών και υπάρχει επίσης μεγάλη μετατόπιση σε ό,τι αφορά τις ε, ισορροπίες ισχύω. Ο Τραμπ έχει διακηρύξει, προεξαγγείλει έναν πόλεμο εμπορίου. Και παράλληλα η κινέζικη πολιτική και η Κινέζικη κινέζικη οδός του μεταξιού ε, καθορίζει τις ε, παγκόσμιες ισορροπίες. Ε, η κατάσταση στη ΣΥΠΑ, η εκλογή ενός δημοχογού που χρησιμοποιεί τον φόβο του κόσμου και τον θωρακίζει με προστατευτισμό αποτελεί σύμβολο των καιρών που επίσης παρατηρείται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν εμφανίστηκε με τον Τραμπ, ούτε πρόκειται να εξαφανιστεί με τον Τραμπ. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να βρούμε κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αντισταθμίσουμε αυτές τις εξελίξεις και αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο μετατόπιση των παραδειγμάτων. Θεωρούμε ότι αυτοί οι εξελίξεις αποτελούν τους αγωνίους λήθους της έκθεσής μου για την παγκοσμιοποίηση και ελπίζουμε ότι με την έκθεση θα μπορέσουμε μεταξύ άλλων να βρούμε στρατηγικές απαντήσεις. Καταφάρ, ό,τι αφορά την κλιματική ατζέντα. Θα πρέπει το θέμα του περιβάλλοντος να μπει εκεί που ήταν αρχικά. Και να ελέγχεται κάθε νέα πολιτική συμφωνία πρώτου τέθει εφαρμογή. Καταρχάς, ύστερα στη συνέχεια, η ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης είναι ένα ζήτημα το οποίο αποτελεί προαπαιτούμενο για τη υποστήριξη των εξωτερικών στρατηγικών. Κατά δεύτερον, η προώθηση της αποδοχής των ευρωπαϊκών πολιτικών ε, στους κόλπους της κοινωνίας των πολιτών με πραγματική διαφάνεια και συμμετοχή και επιτυχή προετοιμασία μίας απάντησης στην παγκοσμιοποίηση με τριθωτικές μεταρρυθμίσεις. Τρίτον, υποστηρίξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων με μια ενιαία και συνεκτική στρατηγική για την συνοχή και τέλος η ταχεία εφαρμογή των μηχανισμών άμυνας, εμπορικής άμυνας, όπως αφορά το dumping, για παράδειγμα. Πέρα από τους βιώσιμους στόχους της χιλιετίας και τους στόχους του αλλαγή του κλίματος, τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αποκριθούν στην μετατόπιση των ισορροπιών και θα πρέπει να υπάρχει και μηχανισμός εφαρμοσιμότητας σε ό,τι αφορά ε, τις συμφωνίες ε, τις εμπορικές και είναι απαραίτητο να υπάρξει και η κοινωνική εταιρική ευθύνη και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσει κάποια μέτρα εσωτερικά. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και σε ό,τι αφορά τι επιχειρήσει και για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των περιβαλλοντικών ε, δικαιωμάτων. Για να επανέλθουμε από εκεί που ξεκινήσαμε, η αλλαγή των παραδειγμάτων λόγω τη κινέζικη και αμερικανικής αλλαγής στρατηγικής, πιστεύω ότι χρειάζεται παρόλα αυτά μια ενισχυμένη συνεργασία με την Ευρασία και μια στεναρή συνεργασία με τα αφρικανικά κράτη. Με τις συμμαχίες αυτές η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ευκαιρία να παραμείνει ένας βασικός ε, παράγοντας στο διεθνές εμπόριο παγκοσμίω. Ευχαριστώ. Sorry, Thank you very much. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σούστερ, τον εισηγητή μας, να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες σκέψεις σε σχέση με το προσχέδιο έκθεσης. Η παγκοσμιοποίηση είναι μια συνεχής διαδικασία και δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις οικονομικές, ε, κοινωνικές, περιβαλλοντικές κλπ. Καλωσορίζουμε το έγγραφο προβληματισμού περί τη θάσευσης της ε, παγκοσμιοποίηση. Ε, η Κομισιόν έχει αναγνωρίσει ότι θα πρέπει. Η παγκοσμιοποίηση δεν έχει μόνο, θετικά, αλλά και αρνητικές, ε, μόνο θετικές, αλλά και αρνητικές επιπτώσεις, ότι θα πρέπει τα ωφέλη να μοιραστούν δίκαια και ότι το εμπόριο είναι ένα μόνο κομμάτι της παγκοσμιοποίησης. αν αποτύχει, εκεί που αποτυχάνει η, δημοκρατία, η οικονομία, αποτυχάνει και η δημοκρατία. Οι, οι πολίτες έχουν όλο και περισσότερη αξιουσία στα χέρια τους, αλλά νιώθουν ότι η δημοκρατία δεν χρησιμεύει τόσο πολύ πια. Η απάντηση στην παγκοσμιοποίηση προφανώς δεν είναι ε, η, το κλείσιμο των συνόρων. Θα, το εμπόριο θα πρέπει να συνεχιστεί, αλλά με κανόνες έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο του κοινωνικού ντάμπινγκ, των υπερβολικά χαμηλών μισθών και τη εκμετάλλευση. Ε, θα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να οθετήσουν βέλτιστες ε, πρακτικές και οι πολυεθνικές θα πρέπει να δώσουν λογαριασμό για τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. Ε, Δεν ε, θα πρέπει οι εκτός οι πολυεθνικές να ε, ρίχνουν το βάρος σε θηγατρικές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαφεύγουν. Το κλείσιμο των συνόρων και ο προστατευτισμός ε, θα, έχει, ε, θα δημιουργήσει ε, ε, το αποτέλεσμα ντόμινο για όλους. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα με διαφάνεια, να, να διασφαλίσουμε στους πολίτες μας ότι είμαστε ισχυροί και να πάρουμε μέτρα ελέγχου και τη θάσευση των δυνάμεων της παγκοσμιοποίησης. Ε, η έκθεση για το εμπορικό κομμάτι της ε, παγκοσμιοποίησης είναι υπερβολικά μικρή σε μέγεθος. Ε, έχουν, έχει όμως σημαντικά σημεία, αλλά δεν αναφέρει το πώς η ε, παγκοσμιοποίηση ευεργετεί τις κοινωνίες. Δεν έχει μόνο αρνητικά σημεία η παγκοσμιοποίηση. Εκεί είναι λίγο αδύναμη η έκθεση. Οι εμπορικές μας συμφωνίες έχουν δεσμεύσει και από τις δύο πλευρές για περιβαλλοντικές, ε, για περιβαλλοντικά στάνταρ, πρόσβαση προς την αγορά, ε, βοηθούν τις αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες ε, οθούνται να υιοθετήσουν χρήσιμες μεταρρυθμίσεις και τους ε, βελτιώνει τη δυνατότητα εξάγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και τι θετικέ πτυχέ τη εμπορική μα πολιτική. Τώρα, το πώ πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα εργαλεία, αυτό είναι το θέμα. Σε ορισμένα σημεία η έκθεση εστιάζεται υπερβολικά στις αδυναμίες δικές μας ή του, του ΠΟΕ δεν πρέπει να εστιάζουμε μόνο σε αδυναμίες. Αντιθέτως, θα πρέπει να δείξουμε πώς μπορούν να βελτιωθούν, να καλυφθούν τα κενά, να ενισχυθούν, να ενισχυθεί το πλαίσιο που, στο οποίο κινούμαστε και το πώς θα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα ή θα συμπληρώσουμε τα εργαλεία μας. Το να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί είναι τμήμα της απάντησης στην διθάσευση της παγκοσμιοποίηση. Το 1 τρίτο του ΑΕΠ μας προέρχεται από ε, διεθνές εμπόριο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν. Ε, η Κομισιόν προσπαθεί να απαντήσει σε αυτές τις προκλήσεις. Είναι σημαντικό αυτό να το αναφέρουμε στην έκθεσή μας. Έχουμε παγκόσμιους στόχους, για παράδειγμα κλιματικούς και βιωσιμότητας. Ε, περιμένω τις διαπραγματεύσεις για να καταλήξουμε σε ένα καλό τελικό αποτέλεσμα. Πρόεδρος. Ποιος Λούνες για την ECR. Ναι εκ μέρους της Emma Μακλάρκιν που δεν είναι δυνατό να παραστεί σήμερα. Και εγώ θα διαβάσω τη δήλωσή της. Όπως αναγνωρίζει ο εισηγητής, οι παγκοσμιοποίηση, οι παγκόσμιες ε, ε, αλυσίδες ε, αξίας έχουν αναμορφώσει το εμπόριο, φέρνουν πιο κοντά τους ανθρώπους και τις αγορές, πολλά τα ευεργετήματα, αλλά δεν θα πρέπει κανένας να μείνει πίσω συμφωνούμε πολλά από όσα λέει η έκθεση, αλλά δυστυχώ διαφωνούμε με ορισμένα, ορισμένες πτυχές της. Ορισμένες προτάσεις, για παράδειγμα, της συγγήτρια. Για παράδειγμα, η συμπερίληψη διατάξεων βιωσιμότητα σε όλα τα κεφάλαια όλων των συμφωνιών με τρίτες χώρες ε, και μηχανισμούς ε, κυρώσεων σε ορισμένα από αυτά το εμπόριο σίγουρα θα πρέπει να στηρίζει την βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά όχι ανάποδα. Οπότε, καλούμε να ακολουθεί μια εμπορική πολιτική με κανόνες που μέσω διεθνών συμβάσεων θα προωθεί τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα και θα στηρίζει τις περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες και συμφωνίες. Δύο σημεία προσθέτως. Αυτή η έκθεση δεν αναφέρεται πλήρως στην δυνατότητα, στην ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνολογίες για να νέες τεχνολογίες για να τη την παγκοσμιοποίηση. Αυτή τη στιγμή ο καθένας μπορεί να ασκεί εμπορική δραστηριότητα από το σαλόν του. Αυτό είναι μια πρόκληση. Ε, ψηφιακή εμπορική στρατηγική χρειάζεται και δεν την έχουμε αναπτύξει ακόμα. Ε, χρήση ιδιαίτερων και νέων τεχνολογιών, τεχνολογιών όπως το blockchain, που δίνουν μάλιστα και μεγαλύτερη ευελιξία και διαφάνεια στο διεθνές εμπορικό σύστημα. Δεύτερον, όπως ανέφερε η κυρία Μόσκα, ή βλέπουμε ότι αναπτύσσονται προστατευτικές τάσεις. Θα πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό, ενισχύοντας τους δεσμούς μας με άλλες ανεπτυσσόμενες οικονομίες, όπως ε, αυτές της Ασίας, του Ειρηνικού, της Λατινικής Αμερικής. Από την άλλη μεριά πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε εξακολουθούν να είναι ο βασικός μας εμπορικός εταίρος Οπότε θα πρέπει να βρούμε μια κοινή προσέγγιση σε διεθνή ζητήματα, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να στηρίξουμε ένα πολυμερές εμπορικό σύστημα που θα στηρίζεται σε κανόνες. Θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες όταν έρθει η ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την συγγήτρια και τους και όδης συγγητές. Σας ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη Ευχαριστώ πολύ. Η ομάδα μου καλωσορίζει το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Σούστερ. Καλώς ορίζουμε την προσέγγιση του, η οποία θεωρούμε ότι αποτυπώνει 100% της προκλήσης στο διεθνές εμπόριο σήμερα. Μία μεγάλη πρόκληση είναι το γεγονός ότι σε γενικέ γραμμέ ο κόσμος ε, είναι αρκετά δυσαρεστημένος με, τα, με τις συνέπειες ε, Τη παγκοσμιοποίηση και κυρίω με τα ωφέλη τη παγκοσμιοποίηση, τα οποία δεν κατανείμονται δικαίω. Αυξάνονται λοιπόν οι ανισότητε και θα πρέπει να βρούμε νέου τρόπου να αντιμετωπίσουμε τι ανισότητε αυτέ και μεταξύ άλλων και με την εμπορική πολιτική. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε λες και δεν συμβαίνει τίποτα με την εμπορική πολιτική και έχουμε πλέον μέχρι το τέλος του 2030 και θα πρέπει να μας καθοδηγούν 17 βιώσιμοι στόχοι και το εμπόριο θα πρέπει να αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της ανοποιημένης προσέγγισης. Δεν μπορούμε να επανέλθουμε λοιπόν στην εμπορική πολιτική παλαιού τύπου και πιστεύω ότι η πολιτική εμπόριο για όλους. Μα πρόεδρε με ακούτε. Με ακούτε γιατί πρέπει να με ακούτε. Πώς θα γίνεται. Ναι, καταλαβαίνω. Κάνετε multitasking, κάνετε πολλά πράγματα. Αλλά Πιστεύω ότι η στρατηγική trade for all της κυρίας Μάλμστρομ είναι μια τέλεια περίπτωση όπου μπορούμε να εντάξουμε την ατζέντα για το 2030. Και σε αυτό το κοινοβούλιο θα πρέπει να βρούμε τρόπο να ανταποκριθούμε σε αυτή την ενοποιημένη ατζέντα στο κοινοβούλιο. Και τώρα έχουμε λοιπόν και την ε, πρόταση του κυρίου Τραμπ στο θέμα αυτό. Προστατευτισμό δεν είναι αυτή η λύση για την Ευρώπη σε καμία περίπτωση, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Θα πρέπει να βρούμε λύσεις όπως και να έχει. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να απαντήσουμε σωστά στην ε, μεταρρύθμιση του εμπορικού συστήματος και του πολυμερούς ε, εμπορικού συστήματος. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να καθορίσει τους κανόνες και όχι να είναι αυτή που τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Ένα καλό παράδειγμα είναι ότι τώρα εισαγάγουμε τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων για όλες τις συμφωνίες πλαίσιο και κυρίως σε ό,τι αφορά το αναδυόμενο εμπορικό, ψηφιακό εμπόριο. Ας είμαστε λοιπόν ενεργοί, ας είμαστε δραστηροί εκ των προτέρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και θεωρείται ηγετική δύναμη σε ό,τι αφορά το περιβάλλον. Θα πρέπει να είμαστε φυσικά ενήμεροι για τις προκλήσεις που είναι τεράστιες σε ό,τι αφορά το διεθνές εμπόριο και τις ε, απόψεις που υπάρχουν ότι είναι αντίθετο με την προστασία του κλίματος. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται πιο πολύ δέσμευση σε ό,τι αφορά την ε, Συμφωνία του Παρισιού σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την εμπορική συμφωνία με την Ιαπωνία. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί και αλλού. Και αυτό αποτελεί μια απόδειξη ότι μπορεί να γίνει ένα τέτοιο συμβιβασμό ε, μεταξύ του εμπορίου και των στόχων για το κλίμα. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιηθεί αυτό ως ένα πρώτο βήμα για μια πιο φιλοδοξή εμπορική πολιτική μεταξύ άλλων και σε πολυμερές επίπεδο για να υπάρξει πλήρη συνοχή σε πολιτικό επίπεδο. Ανέφερε η κυρία Μόσκα ότι θα πρέπει να εργαστούμε για μια υπεύθυνη συμπεριφορά εκ μέρους των επιχειρήσεων. Εδώ λοιπόν πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι πρωτοπόρος δύναμη. Θέλω η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να αναπτύσσει τα πρότυπα του ΑΣΑ για την υπεύθυνη συμπεριφορά των επιχειρήσεων και να προσαρμόσει ανάλογα την νομοθεσία τη Να σα πω ότι στην παρούσα φάση υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη για την ευθύνη αυτή των εταιριών που πολλές είναι οι πρωτοβουλίες και οι νομοθεσίες οι οποίες ε, αναδύονται στα κράτη-μέλη. Εμείς ε, θα πρέπει να φροντίσουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπάρχουν ίσοι ανταγωνισμού και να υπάρξει και μια νομοθεσία για την τέτοια επιμέλεια. Φυσικά είναι σημαντικέ οι πρωτοβουλίε και οι θελούσιε ε, δράσει, αλλά βλέπουμε για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την τριμερή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΠΟΗ και την κυβέρνηση του Μπαγκλαντέ. Αξιέπαινη προσπάθεια, αλλά δεν έχει επιφέρει τις απαραίτητε αλλαγέ για την βελτίωση το βιωτικού επίπεδου και των μισθών στο Μπαγκλαντές, στην Φαντουργία. Άρα έχουν το ρόλο τους ε, οι εθελούς της πρωτοβουλίας, αλλά τώρα πλέον χρειάζεται και μια υποχρεωτική προσέγγιση, πιστεύω. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος, νομίζω ότι το θέμα του Μπαγκλαντές ε, θα πρέπει να το εξετάσουμε, να το παρακολουθήσουμε με προσοχή εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών. Πολλά πρέπει να γίνουν η κυρία Μινέρ και μετά η κυρία Πρόσφα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Έχει... Είναι μεγάλος ο όγκος εργασίας. Ευχαριστώ τον εισηγητή τον κύριο Σούστερ γιατί κάνει αναφορά και στους στόχους ε, ε, της χιλιετίας και στη δέωση επιμέλεια και σε όλα τα στοιχεία τα οποία μας χρειάζονται. Ελπίζω να γίνει πιο φιλοδοξό το σχέδιο να μιλήσω για το εξή. Η εμπορική πολιτική θα πρέπει να εφαρμοστεί με πιο υποχρεωτικό τρόπο σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον και θα πρέπει να πάρουμε λίγο πιο πολύ στα σοβαρά τις μελέτε αντικτύπου. Θα πρέπει να είμαστε στο κοινοβούλιο πιο αυστηροί, να γίνονται μελέτη μελέτε αντικτύπου εγκαίρω, εκ των προτέρων. Και στη συνέχεια τα αποτελέσματά του να τα παίρνουμε σε σοβαρά, γιατί θα είναι κακό και για του πολίτε αλλά και για την εμπιστοσύνη στου πολιτικού από πλευρό των ε, πολιτών. Η αξιολόγηση ITOC. Σε ό,τι αφορά τις ε, ε, πολύ εθνικές εταιρείες που έχουν σημαντικό, α, σημαντική εξουσία. Η ΤΟΚ υπογραμμίζει ότι η παγκοσμιοποίηση ενδεχομένω να οδηγεί σε λιγότερη φτώχεια, αλλά οδηγείται παράλληλα και σε μεγαλύτερη ανισότητα. Εδώ λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα, να δούμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, να δούμε τις ε, συνθήκε της Παγκόσμιας Οργάνωση εργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει, τονίζει ότι αναγνωρίζει ότι οι κυβερνήσει δεν μπορούν να δρασέψουν ε, την παγκοσμιοποίηση, παρόλα αυτά δεν κάνουν ε, καμία πρόταση να γίνουν αλλαγέ. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να ε, εφαρμόσουμε από, να υποχρεωθούν οι επιχειρήσεις να εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες γραμμέ του ΟΑΣΑ. Επίσης, η ITUC υποδεικνύει ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των γενικών διευθύνσεων. Γιατί σε πολλέ περιπτώσει η Επιτροπή έχει αντίθετη δράση. Πολύ περίεργο. Και τέλο, η φοροδιαφυγή που θα πρέπει να αποφευχθεί, να καταπολεμηθεί σε ό,τι αφορά και την ψηφιοποίηση τη εργασία. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε σκληρή δουλειά και κυρίως να βάλουμε και το περιβάλλον ως προτεραιότητα και τις οικονομικές συνέπειες για την απαραίτητη μετάβαση σε ενεργειακό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Εκτός μικροφώνου, δυστυχώς ο Πρόεδρος και ο μιλητής εκτός μικροφώνου. Praising uh, Mrs. Mina for her very lucid contributions, also for her mastery of the English language. I was rather. Κρίμα που δεν άκουσα τα αγγλικά σας. Είναι πολύ καλύτερα από τα δικά μου. Ε, τα μιλάτε τόσο καλά. Ε, ε, πιστεύω ότι η συνεισφορά της κυρίας Χατολά ήταν πολύ σημαντική πολύ πιο ενδιαφέρουσα από ό,τι νομίζει ίδια, από ό,τι καταλαβεί ίδια. Γιατί έβαλε το δάχτυλο στον τύπο των ήλων, στην ρίζα του, των προβλημάτων μας και των συζητήσεών μας. Έτσι όπως το άκουσα εγώ τουλάχιστον και το κατάλαβα. Λέτε ότι ταυτόχρονα ζητάμε και πολλούς καινούριου κανονισμούς για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και για την εφαρμογή της πράσινης ατζέντα. Πολύ σωστά, εντάξει, γι' αυτό ε, ε, εξελέγει η ίδια. Αλλά θέλουμε και περισσότερο εμπόριο και περισσότερες εμπορικές ανταλλαγές. Τελικά θα πρέπει να αποφασίσουμε να σκεφτούμε το εξής. Πόσο μεγάλα είναι τα βάρη τα οποία θέτουμε στο εμπόριο και στη βιομηχανία την κατασκευαστική βιομηχανία, την, κατασκευαστική βιομηχανία αλλά όχι μόνο αυτή. Στα κράτη-μέλη, όσα μείνουν εν πάση περιπτώσει μετά την αποχώρηση της Βρετανίας, προκειμένου να ε, εκπληρώσουμε τους στόχους της κλιματικής ατζέντα, του κλιματικού θεματολογίου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ε, βγαίνουμε χαμένοι ή κερδισμένοι. Εσείς λέτε, Λέτε στην πραγματικότητα ότι είμαστε πράσινοι, οπότε δεν χρειάζεται να παράγουμε αυτοκίνητα στη Γερμανία. Έχετε δικαίωμα να το υποστηρίξετε, αλλά πέστε το ανοιχτά. Θα πρέπει να αναγνωρίσετε τις επιλογές σας και όχι μόνο εσείς, του, στο, οι πράσινοι αλλά και οι υπόλοιποι ε, πρέπει να σταθμίζουμε τα πράγματα και να κάνουμε επιλογές και τις επιλογές μας πρέπει να τις ε, τιμολογούμε να τις κοστολογούμε. Γιατί πολλές από, πολλά από αυτά τα κομμάτια του ρυθμιστικού πλαισίου αποτελούν εμπόδια στο εμπόριο. Μπορείτε να πείτε ότι το αξίζει να τα επιβάλλουμε για τους εξής χίλιους λόγους. Αλλά πέστε το ανοιχτά. Ε, είμαστε, βιαζόμαστε πρόεδρε, σας βλέπω λίγο ανήσυχο. Προσπαθώ να σέβομαι το χρόνο που μου δίδεται κάθε φορά, εν πάση Το άλλο θέμα το οποίο έχω θίξει, το οποίο έθιξα είναι το εξής. Ε, είχα την τιμή να ήμουν μέλο του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακόμα μεγαλύτερη τιμή βέβαια που θα το εγκαταλείψω, με, με, με, με βοήθεια εκατομμυρίων ανθρώπων μεταξύ αυτών και μελών του Κόμματο των εργατικών της Βρετανίας ε, αλλά το θέμα που θέλω να σχολιάσω είναι το εξής συνεχής ε, συνεχ, ε, επανειλημμένη υιοθέτηση νέων κανόνων, νέων νόμων, νέων οδηγιών νέου ρυθμιστικού πλαισίου. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Ήταν η μείωση της ανταγωνιστικότητας της, ελληνικής, της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην παγκόσμια αγορά. Δεν έχω να δώσω απάντηση. Πολύ δε περισσότερο προκειμένου να δώσω μια απάντηση σε τόσο περισμένο χρονικό διάστημα που μου δίδεται. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Ένα τελικό σχόλιο, μια και αναφέρθηκε, αναφέρθηκε τον Μπαγκλαντές. Νομίζω ότι η συζήτηση για τον Μπαγκλαντές παλιότερα ήταν ε, ε, ε ασύμετρη ε, και από πλευρά συμμετεχόντων και από πλευρά απόψεων. Δεν ήταν κανένα μέλος του ΕΛΚ παρόν στη συζήτηση με τον Μπαγκλαντές. Οπότε η συζήτηση δεν ήταν πολύ ε, ισορροπημένη. Θα ζητούσα αυτά τα πράγματα να συζητηθούν και το λέω ταπεινά. Γιατί κάθε αντίδραση έχει και την αντίδρασή της. Αυτό είναι βασικός νόμος της φυσικής, αλλά όχι μόνο της φυσικής και του εμπορίου και της πολιτικής. Πρόεδρος, θα, θα με ενδιαφέρει να δω πώς η Βρετανία θα καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή και πώς θα είναι η, ποια θα είναι η μορφή των εμπορικών συμφωνιών που θα συνάψει αργότερα. Κύριος Ρούμπιχ, ο κύριος Μπούχνερ και η κυρία Χάουταλα. Σα ευχαριστώ κύριε Ρούιμπεχ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συζήτηση αυτή, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ευημερία είναι απόρρια της εργασίας και της παραγωγικότητας και ότι ε, χρειάζονται λοιπόν οι βάσεις αυτές για να μην υπάρχει ε, η φτώχεια που φοβόμαστε. Κοιτάμε λοιπόν την Κίνα όπου έχουμε 400 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν από καθεστώς στόχιας με μια φιλελεύθερη πολιτική. Η Κίνα λοιπόν κατάφερε στον τομέα του εμπορίου να φέρει αμα, ευημερία στον πληθυσμό και αυτό θα συνεχίσει και στο μέλλον. Αυτό που μάθαμε επίσης είναι ότι με τις εξαγωγές αυξάνεται και η ε, αγοραστική δύναμη των πολιτών μας και έτσι αυτή η δύναμη έχει θετικά αποτελέσματα. Και έτσι το κοινωνικό μας λοιπόν σύστημα εξαρτάται από το πώς ε, προχωράει η αγοραστική αυτή δύναμη. Στην Αυστρία, για παράδειγμα, υπάρχει μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη και αυτό συνεπάγεται και καλύτερη ε, συνεισφορά στις ε, εμπορικές, στις, στις φορολογικές υπηρεσίες, στις, φορολογικές, στα έσοδα. σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη των πολιτών μας. Θα πρέπει και αυτή λοιπόν με βιώσιμο τρόπο να αυξάνεται προκειμένου να αυξάνονται και οι εξαγωγές και οι εισαγωγές. Άρα όποιος ε, στρέφεται στον προστατευτισμό τελικά θα καταλήξει σε καθεστώς φτώχειας. Αυτό θέλουμε λοιπόν αυτό και πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε πιο πολύ τους βιώσιμους στόχους της χιλιετίας, ιδιαίτερα στον τομέα των επενδύσεων και της παραγωγής ε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις ε, λιγότερο αναπτυγμένες χώρες να ακολουθήσουμε τον στόχο υπαριθμών 2 γιατί η σίγουρη παραγωγή τροφίμων αποτελεί τον υπαριθμό ένα στόχο γιατί χωρίς ε, τρόφιμα θα φτάσουμε στα τεράστια προβλήματα που διαπιστώνουμε και στην, νότιο, στην Κορέα. Και από την άλλη το νερό είναι ο βιώσιμος στόχος υπερθμών 6, σημαντική σημασία του και αυτού του στόχου. Και τέλος ανανεώσιμες ενέργειες. Χωρίς ενέργεια δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Και Τέλος, να πω ότι αυτό που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι τα, τα σώμαθε υπέρ των υψηλών προτύπων παραγωγής και διαβίωσης σε άλλες χώρες και κοιτάμε τι γίνεται και στην εμπορική πολιτική, την εθνική της κάθε χώρας. Θέλουμε να πετύχουμε λοιπόν μια διεθνή πολιτική η οποία να υλοποιεί τους δικούς μας στόχους, τις δικές μας αρχές, αυτό Από την άλλη επιμένουμε οι διαφωνίες να επιλύονται από εθνικά δικαστηρία. Υπάρχουν πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορά την διευθέντηση αγωγών. Ξέρουμε ε, ότι στο παρελθόν αυτές οι διαφωνίες επιλύονταν με στρατιωτικά μέσα. Ελπίζουμε λοιπόν να μην υπάρχουν τέτοια θέματα πλέον και να ακολουθούνται διαδικασίε οι οποίε θα είναι διαφανεί και θα που επιτρέπουν στι μικρομεσαίε επιχειρήσει να πρόσπιζουν τα δικαιώματά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μπούχνερ, έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λάθος. Ε. Εγώ είχα ζητήσει το λόγο, αλλά ήθελα να ανακοινώσω μία ε, ένα ε, συναγερμό. Δεν είναι συναγερμό όμω για φωτιά για το δικό μα κτίριο. Μάλιστα, λοιπόν, θα πάρω το λόγο. Υπάρχει τάχα μία αντίφαση μεταξύ τη αύξηση ε, του βιωτικού επίπεδου και τη προστασία του κλίματο. Εγώ δεν το πιστεύω Το Πιστεύω ότι ισχύει ακριβώ το ανάποδο. Η Κίνα αναφέρθηκε και η Κίνα πετυχαίνει καλύτερα αποτελέσματα κοιτώντα τι ε, θέσει απασχόληση στον τομέα, για παράδειγμα, των νεώσιμων ε, πήγων ενέργειας. Ε, ε, ακριβώς το αντίθετο ισχύει. σα παρακαλώ λοιπόν α μην υποκρινόμαστε ότι υπάρχει κάποια τέτοια αντίφαση. Και τέλο, η κυρία Χάουτελα λέει ο πρόεδρο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και νομίζω ότι αυτή η επιτροπή θα, κάνει, θα πρέπει να κάνει πιο πολλέ συζητήσει. και σε ευχαριστώ τον κύριο Τάρτμουθ που ξεκινά μια πραγματική συζήτηση. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία καλούμαστε να συζητήσουμε. Να σας πω ότι οι συμπατριδιότητες έχουν πολλούς συνασπισμούς σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και ο πρίγκιπας Κάραλος είναι υπέρ της ε, προστασίας του δικτύου αυτού. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσουμε σε επιχειρήσεις ε, που θέλουν να βελτιώσουν το εργασιακό περιβάλλον, είτε μιλάμε για το μισθό, για τις εργασιακές συνθήκες κτλ. Η δική μου εντύπωση είναι ότι όντω υπάρχουν πιο πολλές, ε, όλο και πιο πολλές επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, που θέλουν να συμμετάσχουν ε, στην αλλαγή αυτή. Αυτές θα πρέπει να υποστηρίξουμε, όχι αυτούς που είναι αναβλητικοί και περιμένουν και θεωρούν ότι το μόνο που έχει σημασία είναι το εμπόριο και τίποτε άλλο. Να σας θέσω την ερώτηση αυτή άμεσα, γιατί είπατε ότι ο κανονισμός αυτός θα οδηγήσει σε μια κατάσταση που ενδεχομένω να μην υπάρξει πλέον βιομηχανία στη Γερμανία. Α, όχι, δεν είπατε κάτι τέτοιο. Είπατε ότι ο κανονισμός αυτός μπορεί να οδηγήσει εκεί. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσει φιλόδοξα πρότυπα για το έτος 2002-2005 τα πρότυπα αυτά καθέστησαν παγκόσμια πρότυπα πολύ γρήγορα και η αμερικανική, η αμερικανή παραγωγή ουσιαστικά επλήχθησαν από την ε, αλλαγή των προτύπων αυτών. Γιατί ο καταναλωτής ήθελε πιο καθαρά αυτοκίνητα και εγώ συνέβαλα το λιθαράκι μου γιατί και εμείς ε, ζητήσαμε, απαιτήσαμε πιο καθαρά καύσιμα για καθαρατρούς κινητήρες. Θα ήθελα λοιπόν κύριε Ντάρτμουθ να σας δώσω αυτή την πρόκληση. Όσο είστε ακόμα μαζί σας και είναι πολύ κρίμα που θα φύγετε, ελπίζω δεν να μην φύγει κανείς, κανένα από τα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου. Ας συζητήσουμε λοιπόν πιο πολύ αυτό το μοντέλο των βιώσιμων επιχειρήσεων. Ας διοργανώσουμε κάτι και από την Επιτροπή μας με την ηγεσία φυσικά του Προέδρου. Φυσικά υπάρχουν ε, αντισταθμίσματα, αλλά γενικά υπάρχει αυτή η προσέγγιση του παλαιού κόσμου και του καινούργιου κόσμου που δεν στέκει. Ε, δεν είμαστε μόνο οι πράσινοι. Νομίζω ότι όλοι α, παρασυρώμαστε από την ε, διάσταση αυτή και όλοι ξέρουμε πώς μπορούμε να δράσουμε διαφορετικά και στο θέμα των πολιτικών. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε πλέον να επιλύουμε ένα θέμα από τη μία και να δημιουργούμε ένα θέμα από την άλλη. Είναι πραγματικά εξαιρετική η χρονική στιγμή να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Και βεβαίω η πραγματική συζήτηση είναι ανταλλάσσουμε επιχειρήματα, και παρακαλώ πείτε και στις ομάδες σας ότι πρέπει να δώσουμε πιστρό χρόνο στην ομάδα, στην Επιτροπή για συζητήσεις και ίσως θα ήταν καλό κάποια θέματα να τα αφήναμε ώστε να είχαμε χρόνο για πραγματική συζήτηση. Ο κύριος Λουκαντικάουλη. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, είναι όντως πολύ μεγάλη η πρόκληση και δύσκολη κατάσταση Μιλάτε για αλλαγές ύφους και επιλογών. Βεβαίως και έχουμε δύο αλλαγές εμείς. Οπωσδήποτε η στρατηγική μας είναι το εμπόριο για όλους και οι αξίες της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας όπως τις ορίζει το θεματολόγιο. Οπωσδήποτε είναι σύμφωνοι με, σύμφωνες με τους στόχους της χιλιετίας. Αυτό άλλωστε ήταν σαφές και όταν υιοθετήθηκε και η ε, πολιτική εξωτερικής δράσης Ευρωπαϊκή Ένωση και με την ε, ομιλία για την κατάσταση τη Ένωση του Juncker πέρσι είδαμε μια μετακύληση του θεματολογίου προς ένα προστατευτισμό που δεν προστατεύει αλλά που εν πάση περιπτώσει πρέπει να ξέρουμε ποια είναι τα στρατηγικά μας ε, συμφέροντα αμοιβαιότητα βέβαια και ενίσχυση δυναμικό των συμφωνιών, των στόχων των συμφωνιών ε, ανοιχτό προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι μόνο μεγάλες κτλ. Ταυτόχρονα, οι ανησυχίε για την ε, παγκοσμιοποίηση δεν έχουν να κάνουν, δεν περιορίζονται μόνο στις ανησυχίες για την οικονομία. Έχουμε μετάλλαξη της κοινωνίας, και σε όρους ψηφιακού εννοείται και από την αντίδραση των κυβερνήσεων θα κριθεί η επιτυχία. Φυσικά πρέπει να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά στη συνεργασία με τα κράτη-μέλη για την πολιτική για την αγορά εργασίας, δεξιότητες, γενικά ανθεκτικότητα της οικονομίας και της κοινωνίας μας στις μεγάλες προκλήσεις, στις ε, εξωτερικές απαντήσεις βεβαίως χρειάζονται τα εργαλεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αξιοποιεί. Ο Επίτροπος σκόμβηση παραδείγματι, με τις προτάσεις για τη φορολογία στον ΩΣΑ, τα ζητήματα για τις μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες, την καταπολέμηση της νομοποίησης παρανομών εσόδων, όλη μας η εξωτερική δράση δηλαδή, αλλά και η εξωτερική έχει μια στρατηγική και κλιματική αλλαγή. Δεν είναι. Δεν αντίκειται στην εμπορική πολιτική κλιματική αλλαγή. Αντιθέτω, θέλουμε να υποστηρίξουμε την μείωση των εκπομπών διοξυκδίου στην μετάβαση προς μια πιο ικανοποιητική οικονομική και εμπορική πολιτική. Ξέρουμε ότι η κλιματική αλλαγή προχωρεί ε, και δεν μπορούμε να την ανατρέψουμε αν δεν αλλάξουμε πολιτική. Αυτό το βλέπουμε συγκεκριμένα και στις συμφωνίες μας με, το, με την Ιαπωνία. Έχουμε παραδείγματι την προεξόφληση της απελευθέρωσης δασμών για πράσινα προϊόντα, πράσινη τεχνολογία, εκεί όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και την πρωτοκαθεδρία και μπορεί να εξασφαλίσει τη δημιουργία πολλών βιώσιμων θέσεων εργασίας ή ανανεώσιμες πηγές, πρόσβαση στο δίκτυο με αμοιβή για αυτόν που παράγει την πράσινη ενέργεια, τον κάθε πολίτη δηλαδή. Όλο και περισσότερο οι πόροι για την κλιματική αλλαγή δηλαδή. Αυτά ευχαριστώ Πρόεδρε και περιμένουμε να δούμε την έκθεση για την περαιτέρω συζήτηση. Κυρία Μόσκα, όχι πολλά σχόλια. Σημειώνω τις ε, προτάσεις των ε, σκιωδών. Πρέπει να υπογραμμίσουμε κάποια από τα στοιχεία που ήδη έχει βάλει ο εισηγητής και φαντάζομαι ότι συνεργάζεται και με τους άλλους σκιώδεις για την ε, ανάπτυξη των σχολείων. Καλώς, ε, τροπολογίες 25 Ιουνίου, 6 το βράδυ. 25 Ιουνίου, 6 το βράδυ. Έγκριση το Σεπτέμβριο. Τελευταίο σημείο. Υπαριθμόν 24. ανταλλαγή απόψεων για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με συμφωνία για την τροποποίηση των εμπορικών πρωτοκόλων τη συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου. Αυτό λοιπόν το πρωτόκολλο. Έχει συζητηθεί πολύ εδώ, στην Επιτροπή και συγκεκριμένα βέβαια σε σχέση με την αντιμετώπιση της Νότιας Σαχάρας και κατόπιν βέβαια της ε, απόφασης του δικαστηρίου το 2016 πρέπει να αλλάξει η αρχική συμφωνία. Έχει οθετήσει λοιπόν την πρόταση το, η Επιτροπή. αρμοδιότητα έχουμε εμείς καθήλυν για τη συζήτηση, αλλά δεν μας ικανοποιούν οι εξελίξεις. Η συζήτηση για τροποποίηση του εμπορικού πρωτοκόλλου έχει προ... ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά ενημέρωση πραγματική δεν έχουμε. Και θυμάμαι και τις συζητήσεις που είχαμε εδώ, στην ίδια μάλιστα αυτή αίθουσα για να ετοιμαστεί ένας κατάλογος των οργανώσεων και εκπροσώπων με τους οποίους έχει έρθει σε επαφή η Επιτροπή σε Μαρόκου για το θέμα της Δυτικής Σαχάρας. Και, αποστολ, και επιστολή στείλαμε και περιμέναμε και να γίνει και συζήτηση στο Συμβούλιο. Και μόνο μετά από πολύ καιρό ήρθε ο κατάλογος. Υπάρχει βέβαια και η θεσμική σύγκρουση τόσο για το εμπόριο σου και για την αλεία. Στο κομμάτι που αφορά το εμπόριο, για την αλεία δεν υπάρχει διαφάνεια. Δεν υπάρχει δημοσιοποίηση δηλαδή του, της συμφωνίας στο, κομμάτι που αφορά τον εξεχρονισμό της αλληλείας. Και αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί η αλληλευτική συμφωνία εκπνέει κάποια στιγμή. Έχει ρητή η μέρα εκπνοής. Κάπου στα μέσα Ιουλίου. Και μου φαίνεται αδιανόητο εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μείνουμε σιωπηλοί εν ώψη μιας προσωρινής εφαρμογή συμφωνίας είτε στην, στον, εμπορικό, στον εμπορικό κλάδο είτε στον αλληλευτικό και να περιοριστούμε μόνο σε μια συνένεση. Γιατί αυτό θα οδηγήσει όχι σε εμπορικό πόλεμο, αλλά σε θεσμικό. Σε θεσμική σύγκρουση δεδομένων και των διοργανικών συνομιλιών. Μεταξύ Επιτροπή Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για την καλύτερη νομοθεσία. Άρα Υπάρχει το κομμάτι της τροποποίησης συμφωνίας που είναι το, του, του εμπορίου και το θεσμικό κομμάτι που έχει να κάνει με τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Εδώ λοιπόν με χαρά δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εισαγωγή και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ο κύριος Φερνάντο Περόντε Πινόκ έχει το λόγο. Όχι, με συγχωρείτε, μια μικρή σύγχυση στις επιδογραμματίες. Θα ομιλήσει η Σαμπίρια Χέντσλε πρώτη, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι κύριε και κύριοι. Καταρχάς να σας συστηθώ, γιατί είμαι και καινούργια στην Επιτροπή. Σαμπίρε Χένσλερ ονομάζομαι και είμαι επικεφαλής διευθυντρία για τις διεθνείς σχέσεις στα θέματα Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνιακής Ένωσης. Και κληρονόμησα το φάκελο αυτό από 1η Φεβρουαρίου 2018. Έχω λοιπόν τη χαρά σήμερα να βρίσκομαι εδώ μαζί σας για να κάνουμε την ανταλλαγή αυτή απόψεων μαζί σας. Και πρόταση λοιπόν σε ό,τι αφορά την διεύρυνση των ε, δασμολογικών ρυθμίσεων για τη Δυτική Σαχάρα. Η πρότασή μα ε, τροπολογεί τα πρωτόκολλα 1 και 4 τη Συμφωνία Σύνδεση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μαρόκο. Προκειμένου να συμμορφωθούμε με τι απαιτήσει ε, της τη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Δεκεμβρίου του 2016. Ο στόχος μας είναι διπτό. Πρώτον, προτείνουμε μια νομική βάση για να δώσουμε προτιμησιακό τελωνιακό καθεστώ ε, σε προϊόντα της Δυτικής Σαχάρα. Αυτές οι προτιμήσεις ε, είναι παρόμοιες με αυτές που χορηγούνται στο Μαρόκο μέσω της ε, τρέχουσας συμφωνίας σύνδεσης με το Μαρόκο και δεύτερος στόχος μας εξασφαλίζοντας να εξασφαλίσουμε ότι οι εξαγωγές προϊόντων της Δυτικής Σαχάρας θα μέσω των προτιμήσεων θα βοηθήσουν στην βελτίωση της ευημερία των κατοίκων της Δυτικής Σαχάρας και στην σταθεροποίηση της περιοχής της Δυτικής Αφρικής, του Δυτικού Μαγκρέπ. Ε, ε έχουμε πάρει προτάσεις από άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από την Επίσης Εξωτερικών Υποθέσεων, ε, Εξωτερικής Δράσης. Ε, το έγγραφο αυτό περιγράφει το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων που έγιναν με ένα αριθμό φορέων οργανώσεων ε, και ομάδων της Δυτικής Σαχάρας, μεταξύ αυτών και το μέτωπο Πολυσάριο. Και δεύτερον, περιγράφουμε τα ωφέλη που θα προκύψουν για την οικονομία και τον πληθυσμό της Δυτικής ε, Σαχάρας. Να υπογραμμίσω τα έξι βασικά σημεία κλειδιά, τα οποία θα πρέπει να έχετε υπόψη για την πρότασή μας. Πρώτον, σεβασμός του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. το σχέδιο συμφωνίας ε, συνάδει πλήρως με τις απαιτήσεις του, ευρωπαϊκού, του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως περιγράφηκαν στην απόφαση του 2016. Βασίζονται οι προτάσει μα σε μια ευρεία διαβούλευση με όλους τους εμπλεκομένους, συμπεριλαμβανομένου και του μετόπου Πολυσάριου, όπω είπα, που απέρριψε την πρόταση γιατί θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαπραγματευτεί μαζί τους και όχι με το Μαρόκο. Επίσης, βασίζεται σε, μια, σε βάθος ανάλυση των κοινωνικο-οικονομικών ωφελών που θα προκύψουν από τις τελωνιακές προτιμήσεις για τον πληθυσμό και την οικονομία της Δυτικής Σαχάρας. Δεύτερο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι το καθεστώς της ε, Δυτικής Σαχάρας στη διαδικασία του ΟΗΕ αναφέρεται σαφώς στην πρότασή μας ότι η, το προσχέδιο συμφωνίας δεν προκαταβάλει ε, την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά το καθεστώς της Δυτικής Σαχάρας, ούτε και αποτελεί έμεση αναγνώριση της κυριαρχίας του Μαρόκου στην ε, επικράτεια της Δυτικής Σαχάρας. Η πρότασή μας στηρίζει ρητά την διαδικασία του ΟΗΕ προκειμένου να βρεθεί μια οριστική πολιτική λύση στο θέμα της Δυτικής Σαχάρας. Στηρίζουμε πλήρως τις ε, νέες ε, πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΕΕ να βρεθεί μια πολιτική λύση σε αυτή τη μακρόχρονη διένεξη. Η, ε, είπατε εκπρόσωπος κυρία Μογκερίνη έχει συναντηθεί δύο φορές με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και με τον απεσταλμένο του ΟΗΕ στη Δυτική Σαχάρα και στηρίζει τι προσπαθίε του. Τρίτο σημείο. Η, τα ωφέλη για τον ντόπιο πληθυσμό. Η έκθεση για αυτά βασίζεται στην ανάλυση δεδομένων που έχουμε στα χέρια μας και προβολή αυτών στο μέλλον. Σε γενικέ γραμμέ υπάρχουν ενδείξεις ότι η χορήγηση προτιμησιακού καθεστώτος στα προϊόντα της Δυτικής Σαχάρας θα δώσει πολύ ε, σημαντική όθηση στις ε, εξαγωγές, στην οικονομία και στις επενδύσεις σε αυτή τη χώρα. Ε, αν δεν γίνουν δεκτές, ε, η, χώρα, η περιοχή θα οδηγηθεί σε οικονομική αστάθεια. Ε, τα περισσότερα βιομηχανικά προϊόντα και γεωρικά προϊόντα της Δυτικής Σαχάρας θα εισάγονται με βάση αυτές τις προτάσεις χωρίς δασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, τα προϊόντα στη Δυτική Σαχάρα θα έχουν τι ίδιε προτιμήσει, το ίδιο προτιμησιακό καθεστώ με αυτά του Μαρόκου. Αν δεν γίνουν δεκτέ αυτέ οι προτιμήσει, οι εξαγωγέ από την Δυτική Αφρική θα είναι σε μειονεκτούσα σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τις εξαγωγές άλλων χωρών της ίδιας περιοχής, οι οποίες έχουν υπογράψει ε, ή εμπορικές συμφωνίες ή έχουν ενταχθεί στο γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων. Οι διαβουλεύσει με τους φορείς της Δυτικής Αχάρας σε γενικές γραμμέ, δείχνουν ότι υπάρχει επιθυμία να επωφεληθούν των ε, προτιμησιακών ε, ε, ε, προτάσεων. Ο συνάδελφός μου θα σας ενημερώσει σε λίγο γι' αυτό. Τέσταρτο στοιχείο που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας είναι η ίδια η διαβούλευση που έγινε. Ο συνάδελφο από την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, ε, ο κ. Πικέ, θα σα δώσει περισσότερε λεπτομέρειε. Να σα πω όμω εγώ δύο πράγματα γι' αυτό. Ε, διαβουλευθήκαμε με τον το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό φορέων. Μεταξύ αυτών, το μέτωπο Πολυσάριο. Σε γενικέ γραμμέ, η διαβούλευση απέδειξε ότι το σχέδιο συμφωνίας χέρι ευρεία στήριξης. Οι, οι λόγοι πίσω από τις οποιασδήποτε αντιρρήσεις και οποιαδήποτε απόρριψη δεν έχουν άμεση σχέση με την ίδια τη συμφωνία και τον αντικτυπό της. Ε, έχουν σχέση πιο πολύ με την άποψη ε, των συγκεκριμένων ομιλητών μα σε ό,τι αφορά το καθεστώς της Δυτικής Σαχάρα και τη διαδικασία του ΟΗΕ. Οι αντιρρήσει τους βασίζονται δηλαδή σε πολιτικά πιο πολύ επιχειρήματα και όχι κοινωνικο-οικονομικά. Αυτό όμως που συζητούμε εδώ σήμερα είναι ένα όργανο εμπορικής, ένα εργαλείο πολιτικής, εμπορικής πολιτικής. Ε, το εντυπωσιακό είναι ότι οι ομάδες που αρνούνται την επέκταση των, του προτιμησιακού καθεστώτος στη Δυτική Σαχάρα δεν εντοπίζουν κανόνας είδου αρνητική ενδεχόμενη επίδραση, επίπτωση αυτού του συστήματος που προτείνουμε. Για μας ε, δεν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στο να στηρίξουμε την οικονομική και εμπορική ανάπτυξη στη Δυτική Σαχάρα με την ταυτόχρονη στήριξη των ε, προσπαθειών ε, της Δυτικής Σαχάρας για την ε, απόκτηση συγκεκριμένου καθεστώτος κυριαρχίας. Το αντίθετο, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο τις προσπάθειες του ΟΗΕ. Πέμπτο σημείο. Δεν προτείνουμε καμία αλλαγή στις συνθήκες πρόσβασης αγορές. Η συμφωνία, η προτιμησιακή συμφωνία δεν θα αλλάξει την κατάσταση των αγορών σε σχέση με πριν. Δεν δημιουργούνται καινούριε προτιμήσεις δηλαδή. Από την ε, απόφαση του Ευρωπαϊκού Αστηρίου και μετά ε, τα, οι εξαγωγέ τη ε, Δυτική Αχάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Όμω με τι προτάσει μα αυτοί οι δασμοί θα μηδενιστούν. Έκτο σημείο. Η εταιρική σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση Μαρόκο. Η... Το σχέδιο συμφωνία είναι σημαντικό για να αναπτυχθεί αυτή η εταιρική συμφωνία. Το Μαρόκο είναι χώρα κλειδί στην στρατηγική γειτονία μας. Και είναι πολύ σημαντικός παράγοντας ε, σε πολλούς τομεί όπως η μετανάστευση, ο οικονομικός, ο κοινωνικός, ο εμπορικό κλπ. Και αυτή η πρότασή μα θα παίξει σοβαρό ρόλο στην ενίσχυση των σχέσεών μας με το Μαρόκο. Να σας πω και δύο-τρία πράγματα για το περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε. Προτείνουμε η συμφωνία συναυθεί με το βασίλειο του Μαρόκου, διότι είναι ο μόνος πρακτικός τρόπος να παράσχουμε προτιμησιακή ε, μεταχείριση για τα προϊόντα της Δυτικής Σαχάρας. Υπό τις τρέχουσες συνθήκες δεν υπάρχουν φορείς στη Δυτική Σαχάρα που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την εφαρμογή αυτού του συστήματος. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και την επιβεβαίωση της προέλευσης των προϊόντων και την απαραίτητη συνεργασία με τις τελωνιακές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερο σημείο. Η, το σχέδιο συμφωνίας περιλαμβάνει δέσμευση και από τις δύο πλευρές περί ανταλλαγής πληροφοριών τουλάχιστον άπαξ ετησίως. Αυτή η ρήτρα θα μας επιτρέψει να αξιολογούμε τακτικά και ενδεχομένως να βελτιώσουμε τη συμφωνία και τον αντίκτυπό της στην Δυτική Σαχάρα. Και τρίτο σημείο, η Κομισιόν δεν προτείνει προσωρινή εφαρμογή, το είπατε στην εισαγωγή σας, αναμένουμε ότι η συμφωνία θα συναυθεί γρήγορα προκειμένου να ωφεληθεί ο λαός της Δυτικής Σαχάρας και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια, η νομική ασφάλεια και η σταθερότητα. Τώρα να δώσω το λόγο στον συναδελφό μου τον κύριο Ντεπίνινγκ που θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα ωφέλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε Σαμπίνε και θα παρουσιάσω τα βασικότερα στοιχεία της έκθεσης. Σε πέντε λεπτά, αν μπορείτε, λέει ο και σε λιγότερο. Το πρώτο σημείο, λοιπόν, είναι ότι βασιστήκαμε σε μία ποικιλία πηγών. Εσωτερικές πηγές, δημοσιεύσεις, ευρωπαϊκές ε, αντιπροσωπείες, διαβουλεύσεις με τα ενδιαφέρομενα μέτρα, μέρη, ε, μαροκινούς ομολόγους και σε ό,τι αφορά λοιπόν την οικονομία της Δυτικής ε, Σαχάρας διαπιστώνουμε ότι βασιζόμαστε κυρίως ε, στην Αλία και στα Μιλάμε για πάνω από 6.000 εκμεταλλεύσεις ε, και απασχολούνται εκεί 35.000 άτομα περίπου. Και μιλάμε κυρίως για ντομάτες, πεπόνια, 65 εκατομμύρια ευρώ περίπου στην αξία τους. Υπάρχουν και κάποια παραδοσιακά έτη, τα οποία όμως έχουν μικρότερη αξία. Αυτά στη Ρωσία εξαγάγονται κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διοχετεύονται και στην ιστορική αγορά στο Μαρόκο. Οι προοπτικές λοιπόν του τομέα της γεωργίας είναι οι εξή. Υπάρχουν σχέδια επέκτασης της παραγωγής και των εκτάσεων που καλλιεργούνται Κάποια στοιχεία μιλάνε και για πενταπλασιασμό των εκτάσεων αυτών για δημιουργία θέσεων εργασία που φτάνουν μέχρι και τι 65.000. Αυτά είναι σχέδια φυσικά. Υπάρχει λοιπόν αντικτύπω και στου υδάτινου πόρου, γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τις νέες τεχνολογίες για την αξιοποίηση των φυσικών πόρων σε ό,τι αφορά τα προϊόντα της αλίας. Εδώ είναι σημαντικό να υπάρχει σωστός ορισμός ε, του αλευτικού προϊόντος. Μεταποίηση των ε, αλευτικών προϊόντων σε ε, επιχειρήσεις που βρισκόνται στη Βετική Σαχαρά για ψάρια τα οποία έχουν είτε αλλιευθεί στη Σαχάρα και στη Βετική Σαχάρα ή στα χωρικά υδατά του Μαρόκο ή από ευρωπαϊκά σκάφη και μαροκινά σκάφη στα διεθνή υδατά. Έχουμε πάνω από 100 εγκαταστάσεις ε, που έχουν την ε, άδεια να μεταποιούν τέτοια προϊόντα και να τα εξαγάγουν στην Ευρώπη. Μιλάμε για μια όγκο παραγωγή σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ. Τα μισά εξ αυτών εξαρτώνται από τις ε, εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τώρα τα φωσφορούχα, δεν έχουμε στοιχεία στην παρούσα φάση. Υπάρχει αγορά για τα λοιπάσματα και ιδιαίτερα τις εκτιμήσεις που ανέρχονται γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρον λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια θα ήταν λοιπόν η αντίκτυπος μιας συμφωνίας, σύμφωνα με την ανάλυση μας. Θα ε, έδινε δυνατότητα εξαγωγής αλληλευτικών προϊόντων υπό προνομιακούς όρους ε, μετά την διακοπή των προνομιών τον ε, Δεκέμβριο του 2016. Επίσης, θα διευκόλυνε τις επενδύσεις στους κλάδους αυτούς. Και ποιος ήταν ο αντίκτυπος του να μην επιτευχθεί συμφωνία. Καταρχάς, οι εξαγωγές από τη Βυτική Σαχάρα θα βρισκόντουσαν αυτόματα σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τις εξαγωγές από το Μαρόκο και από τις γειτονικές χώρες, γιατί δεν θα υπήρχαν εμπορικές προτιμήσεις. Θα υπήρχε αβεβαιότητα φυσικά στους κλάδους αυτούς, αυτό θα είχε αντικτύπω και στις θέσεις απασχόλησης και στην οικονομική δραστηριότητα, γιατί αυτές οι προτιμήσεις έχουν σημαντική αξία, ιδιαίτερα στα γεωργικά προϊόντα και σε κάποια λευτικά προϊόντα για τα οποία οι δασμοί είναι υψηλή, πιο υψηλοί. Επίσης, θα μπορούσε να διακυβεύσει και τις ε, μελλοντικέ επενδύσεις στον κλάδο αυτών και των αλευτικών προϊόντων και των φωσφορικών αλάτων. Και τέλος, θα σήμαινε τη μετατόπιση της οικονομικής δραστηριότητας από τη Δυτική Σαχάρα, η παραγωγή, οι επενδύσεις θα μεταφέρονταν σε άλλες περιοχές που έχουν προτιμήσεις, το οποίο δεν θα σήμαινε απαραίτητα ε, τις γειτονικέ περιοχές του Μαρόκο για τις μειονεκτούσες περιοχές. Ευχαριστώ. Βινσάν Πικέ, παρακαλώ. Ή Βίνσεν Πίκετ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Θα περιοριστώ στα κύρια θέματα της ε, πολιτικής, της εξωτερικής πολιτικής ε, που αφορούν αυτή την πρόταση και κυρίως την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και τις συνέπειες που απορρέουν από αυτήν. Καταρχάς. Και μετά θα εστιαστώ στις διαβουλεύσεις. Πρώτον, προφανώς είναι δεσμευτική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για όλους μας και η πρόταση που βλέπετε αντικατοπτρίζει πλήρη εφαρμογή της. Τι μας λέει το δικαστήριο. Στην απόφαση για τη γεωργία, αλλά λίγο πολύ το ίδιο είναι ή πολύ πολύ το ίδιο είναι και αυτό που λέει για την αλία. Λίγο νωρίτερα ήρθε αυτή. Ότι είναι ισχυρές οι συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου αλλά ελείψει ειδική ρητής αναφοράς στο, ε, στα αυτόνομα εδάφη της Δυτικής Σαχάρας δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στην περιοχή αυτή. Το δικαστήριο δεν λέει ότι είναι αδύνατον να συμπεριληφθεί και να καλυφθεί και η Δυτική Σαχάρα σε μια συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Μαρόκο. Λέει όμως ότι εάν υπήρχε ο σκοπός να συμπεριληφθεί η περιοχή της Δυτικής Σαχάρας σε αυτή τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου θα έπρεπε να έχει γίνει ειδική μνήα και να προβλεφθούν ειδικέ συνθήκες. Ποιε είναι αυτές οι συνθήκες. Πρώτα απ' όλα, μιλήματα σχετικά με το διεθνές δίκαιο. Την διαδικασία δηλαδή εν εξελίξει επίπεδο ΟΗΕ για τη Δυτική Σαχάρα, μια διαδικασία που έχει ήδη ιστορία δεκαετιών που στόχο έχει να καταλήξει στον προσδιορισμό του τελικού καθεστώτος ε, για την περιοχή αυτή. Ε, υπογραμμίζεται και επαναλαμβάνεται το σύνολο των δεσμεύσεων και αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το δικαστήριο. Δηλαδή λέει ότι ό,τι και να γίνει στο πλαίσιο αυτής της ε, συμφωνίας ε, θα γίνεται πάντα με επιφύλαξη αυτής της ε, διαπραγμάτευσης, της διαβούλευσης επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Δεν πρέπει δηλαδή να βρεθεί σε πιο προνομιούχο ή λιγότερο προνομιούχο θέση η μία ή μια πολύ σοβαρή προσπάθεια από το δικαστήριο να μείνει ουδέτερο και αναφέρεται ξεκάθαρα στο ε, με ποιο τρόπο πρέπει ή μπορεί να υπάρξει κάλυψη της Συμφωνίας ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου για τη Δυτική Σαχάρα και απευθύνει έκκληση ξεκάθαρα στις δύο πλευρές να συνεχίσουν τη διαδικασία με στόχο την εξέβρεση μιας αμοιβαία αποδεκτής και βιώσιμης λύσης στο ζήτημα με ε, τελικά μια συνταγματική τάξη και κάλυψη της ε, περιοχής αυτής μέσα από τη διαδικασία των Ηνωμένων Αυτά λοιπόν. Εμείς διατυπώσαμε τη βασική αρχή της ε, συμβατότητας με το Διεθνές Δίκαιο, υποτασσόμενη σε αυτή την αποφάση του δικαστηρίου. Και τώρα στο δεύτερο ζήτημα, που έχει να κάνει με, την, ε, με το σκεπτικό της απόφασης, σε σχέση με τη Δυτική Σαχάρα. Πιο περίπλοκο ζήτημα βέβαια. Και βέβαια σχετικό με το ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με τη Δυτική Σαχάρα. Δηλαδή καταλήγουμε σε μια ατελή κατάσταση, μια πολιτική και σταγματική κατάληξη, κατάσταση που δεν έχει ολοκληρωθεί σε σχέση με τη Δυτική Σαχάρα. Άρα τι γίνεται, σε ποιον θα μιλάμε, με ποιον θα επικοινωνούμε, αν χρειάζεται να στήσουμε τη γνώμη των ε, ανθρώπων στη Δυτική Σαχάρα. Προκειμένου λοιπόν να κάνουμε σεβαστή τη διαδικασία των ΗΠΑ επιλέξαμε να απευθυνθούμε σε πληθώρα αντισυμβαλωμένων. Αφενός μεν επίσημη, γιατί είναι τρί, τρίπτυχο αυτό στο οποίο απευθυνόμαστε, αφενός μεν τους επίσημα εκλεγμένους ε, και εκπροσώπους της Δυτικής Σαχάρας στο Μαρόκο, στη Βουλή, στις, στα περιφερειακά συμβούλια, περιφερειακά επιμελητήρια περί τους 120 συγκεκριμένα. Έχω δει τον κατάλογο των ονομάτων. Και είναι Σαχράουι στην πραγματικότητα. Προέρχονται λοιπόν από την ε, έχουν την εθνοτική καταγωγή των Σαχράου και έχουν συμπεριληφθεί σε αυτόν τον κατάλογο του πρώτου, τριπτύχου, του πρώτου του σκέλους του τριπτύχου. Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με διαβουλεύσεις με το μέτωπο Πολυσάριο, συνάντηση που έλαβε χώρα εδώ στις Βρυξέλλες και από την οποία με ένα-δύο θέματα βέβαια στην ημερήσια διατάξη, το 90% ε, των ε, ανταλλαγών είχε να κάνει με την γεωργία. Εγώ προείδρευσα τη συνεδρίαση και ρώτησα συγκεκριμένα εάν υποστηρίζει την προσέγγιση αυτή το μέτωπο Πολυσάριο. Η απάντηση που έλαβα ήταν αρνητική για λόγους πρωταρχικά πολιτικούς που έχουν να κάνουν με, την, ε, με τον πολιτικό συλλογισμό που ακολουθεί το μέτωπο Πολυσάριο, το οποίο ευθύ μπορούν να σα εξηγήσουν καλύτερα, πάντως όχι εγώ. Θα είδατε ίσως και κάποια άρθρα στον τύπο από τα οποία αντικατοπτρίζεται αυτή η αρνητική στάση του Πολυσάριο. Και το τρίτο, το τρίτο σκέλος έχει να κάνει με ε, επικοινωνία με μια σειρά από φορείς που δεν έχουν ε, θεσμικό χαρακτήρα κρατικό Επομένω, έχουμε να κάνουμε κυβερνητικέ οργανώσει, κοινωνικο-οικονομικά σώματα, εκπροσώπου πολιτών κτλ. Συναντήσεις είχα στο Ραμπάτ, ορισμένες και στις Βρυξέλλες, όπου και πάλι η ερώτησή μου ήταν πάντα αν συμφωνούν με την προσέγγιση και η απάντηση που ήταν πάντα θετική. Κάποιοι από τους ε, ανθρώπους με τους οποίους επικοινωνήσαμε, από τους φορείς με τους οποίους επικοινωνήσαμε, δεν δέχτηκαν την πρόσκληση, δυστυχώς, αλλά υπήρξε από άλλους θετική ανταπόκριση. Και κάτι ακόμη, για να ολοκληρώσω, θα ήθελα να τονίσω ότι με αυτή την τόσο ε, ανοιχτή και συμπεριληπτική ε, ε, προσέγγιση, ανοιχτή προς όλους δηλαδή, νομίζω ότι και υλοποιούμε αυτό που ανέφερε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νωρίτερα, ότι απευθυνόμαστε στο λαό της Δυτικής Σαχάρας. Με αυτούς επικοινωνούμε προκειμένου να αξιολογήσουμε και να εξασφαλίσουμε την ε, συνένεση για να προαχθεί αυτή η συμφωνία. Ευχαριστώ. Πρώτη για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την πρότασή σα την πρόταση Κομισιόν. Οπότε, προς το παρόν, βασικά μόνο ερωτήσεις και όχι μακροσκελείς τοποθετήσει. Θα δώσω 1,5 λεπτό στο κάθε συνάδελφο. Παρακαλώ πολύ να είστε ακριβείς και ολιγόλογοι. Οι συντονιστές επίσης αποφάσισαν χτες αφενός να υποβάλουμε ένα ψήφισμα στη διαδικασία σύμφωνη γνώμη, να αναφέρουν ποια είναι οι δικέ μα απαιτήσει, οι δικοί μα όροι. Και δεύτερον, να ζητήσουν να γίνει μια ερευνητική αποστολή στη Δυτική Σαχάρα. Για να αποκτήσουμε η ίδια εικόνα. 1,5 λεπτό λοιπόν στον καθένα ερωτήσεις και εν συντομία παρακαλώ. Πρώτα ο λόγος στην κυρία Λαλόν, την εισηγήτρια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Χαίρομαι που γίνεται αυτή η ανταλλαγή απόψεων σήμερα με την Κομισιόν. Μία εβδομάδα αφότου το κοινοβούλιο μας ε, έλαβε την ανταλλαγή επιστολών για τις διαπραγματεύσεις από τον πρωτοκόλλο 1 και 4 Ευχαριστούμε που η Κομισιόν μας παρουσίασε την εργασία της. Δεν θα είναι η μοναδική ευκαιρία που θα έχουμε. Και για αυτή τη συμφωνία και για τη συμφωνία Αλίας, το διακύβευμα δεν είναι μόνο οικονομικό και εμπορικό. Είναι πολιτικό και διπλωματικό πάνω απ' όλα. Και γι' αυτό θέλω να τοποθετηθώ. Η η διαμάχη γύρω από τη Δυτική Αφρική αποκαλείται παγωμένη διαμάχη. Η ίδια επικράτεια ε, διεκδικείται από το, με το Πολυσάριο και από το Μαρόκο. Αυτή τη στιγμή ε, η συμφωνία ε, έχει βέβαια ως στόχο ε, να ωφεληθούν όσοι ζουν στη Δυτική Σαχάρα και μάλιστα με τον ίδιο τρόπο με αυτόν που ωφελούνται οι κάτοικοι του Μαρόκο από τις εξαγωγές τους. Αλλά μπορεί να ειδωθεί ως μοχλός στην ειρηνευτική διαδικασία ανάμεσα στο μέτωπο Πολυσάριο και στο Μαρόκο. Αυτό είναι για μένα η ουσία του θέματος που είναι πολιτικό. Τώρα, από την άλλη μεριά, όλοι συμφωνούμε να στηρίξουμε τις προσπάθειες του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει εδώ. Μόνο αυτές οι προσπάθειες ε, είναι θεμητές. Τώρα, για να ξαναξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, πρέπει ο καθένας να κάνει ό,τι του αντιστοιχεί. Θα πρέπει κάπως να κινηθούν τα πράγματα. Το Μαρόκο και το μέτωπο Πολυσάριο, χωρί προϋποθέσεις, ε, χωρί όρου να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Τέλειωσα, εισηγήτρια είμαι. πώ να προλάβω κύριε Πρόεδρε. Τι μου δίνετε, δύο λεπτά. Θα συνεχίσω. Θα ήθελα να στηρίξω την πρόταση της Αλγερίας στο Μαρόκο να στηριχθεί για να διοργανώσει το ε, Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Ορισμένοι πολιτικοί Αλγερινοί όπως ο Σαϊτ Σαϊντή έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ Μαρόκου και Αλγερίας έτσι ώστε να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση για τη Δυτική Σαχάρα υπό την αιγίδα του απεσταλμένου του ΟΗΕ. Αν αυτό το θέμα μας βοηθήσει να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση θα χαρώ ιδιαίτερα. <laughs> Merci beaucoup. C'est quand même un peu sévère. Yeah, but... Πρόεδρος. Είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων, κύριε Λαλόντ. Μόλις τώρα μας παρουσίασε την πρόταση η Κομισιόν. Για ερωτήσεις σας δίνω το λόγο, όχι για τοποθετήσεις. Θα ξαναγίνει συζήτηση. Θα έχουμε ευκαιρίες να προσθέσετε την άποψή σας. Μην ανησυχείτε. Και η συγκήτρια θα, πάει, θα έχει αρκετό χρόνο για να, παρουσιάσει το ψήφισμά της. Σήμερα επικεντρωνόμαστε σε, στην παρουσίαση της πρότασης. Ε, ο κ. Τσίκο για το ΕΛΚ. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ακολουθώ τις, τις υποδείξεις σας. Επομένως, εστιάζομαι σε ερωτήσεις. Ωστόσο, πιστεύω ότι πέραν όλων των σημαντικών βεβαίω θεμάτων, πρέπει να εστιαστούμε στο εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιλέξει την καταλληλότερη μέθοδο προσέγγισης και με βάση και τις ενδείξεις και υποδείξεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πρέπει να καταλάβουμε δηλαδή εάν αυτές οι ακροάσεις που οργανώθηκαν και ε, πραγματοποιήθηκαν είναι συμβατές με τις υποδείξεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ιδάλλως, αντιμετωπίζουμε και πάλι τον κίνδυνο των προσφυγών και της αμφισβήτησης της νομιμότητας της επικαιροποίησης. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό, λεπτό και ευαίσθητο το θέμα συμφωνώντας πάντα με το περιεχόμενο του ψηφίσματος και του τρόπου με τον οποίο και του ρόλου που έχει τον, του αυτόνομου αλλά και του πρωταγωνιστικού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να κάνει τις δικές του τις αξιολογήσεις, θα πρότεινα να αναθέσουμε στις νομικές μας υπηρεσίες να μας πούν να κάνουν μια εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει το ζήτημα ή πώς θεωρούν ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίζει το ζήτημα. Ευχαριστώ, Εμμανουέλ Μοχέλα, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ. Προήμιο. Μεταξύ μας συζήτηση δεν τίθεται ως προς το τι θέση έχουμε για την Δυτική Σαχάρα, γιατί προφανώς έχουμε πολύ διαφορετικές θέσεις. Εγώ συγκεκριμένα μάλλον προσεγγίζω τις θέσεις της γαλλικής διπλωματίας, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημά μας. Το θέμα είναι πώς μπορούμε και να κάνουμε σεβαστή την απόφαση του δικαστηρίου και ταυτόχρονα να διαφυλάξουμε τις στρατηγικές μας σχέσεις με το Μαρόκο που είναι τόσο σημαντικέ. Τα προϊόντα που προέρχονται από τη Δυτική Σαχάρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούν πλέον να λαμβάνουν τι ε, δασμολογικέ προτιμήσει. Παράδοξο βέβαια για περιοχή που θα θέλαμε να υποστηρίξουμε το θέμα είναι πρέπει να την αποκλείσουμε από κάθε συμφωνία, προφανώ όχι. Για το περιεχόμενο, συνένεση των πολιτών, των ε, κατοίκων θεωρείτε ότι έχετε κάνει αρκετά θα μπορούσε να υπάρχει κάτι περισσότερο πιο βιώσιμο και πιο ουσιαστικό στην επικοινωνία δεύτερον όφελος για την περιοχή την ίδια ή τοπικό όφελος δηλαδή το να πούμε μόνο αλία μόνο γεωργία δηλαδή επαγγέλματα που η απασχόληση που δεν μπορεί να μετατοπιστεί αρκεί αυτό σαν επιχείρημα ή μήπως πρέπει να κοιτάξουμε να ανοίξουμε λίγο περισσότερο την ε, ε, βεντάλια και σε αυτό που είπε και ο Μπερτράν, υπάρχει ένα ζήτημα μεθόδου. Νόμιζα ότι αυτό ήταν και το δόγμα που ακολουθούν οι γενικά τα θεσμικά όργανα. Δεν, δίνεται δεν δίνεται να γίνει προσωρινή συμφωνία χωρίς συνένεση του Κοινοβουλίου. Επομένως, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σε διαπραγματεύσεις αδιαφανείς, ενημέρωση ελιπέστατη, πληροφορίες που μας λείπουν, παρότι όλοι θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η εταιρική σχέση, στρατηγική σημασία εταιρική σχέση με το Μαρόκο. Και σταματώ εδώ. Κύριος Μπούχνερ, πράσινε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήδη προβλήματα μου γεννά ο τίτλος όταν, λέτε για, όταν μιλάτε για population, πληθυσμό στην έκθεση. Πώς λοιπόν μπορεί να συγκεραστεί αυτό με την απόφαση του δικαστηρίου, γιατί το δικαστήριο μιλάει για λαό των Σαχράουι και όχι για πληθυσμό της Δυτικής Σαχάρας. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και το είπατε σε τελευταία ανάλυση, αναφέρθηκε ο υπήν, με κάποιους συνεργάτες ε, συνεργαζόμενους από τους Σαχράουι με τις αρχές του Μαρόκου ήρθατε σε επαφή. Με κάποιες ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις από τις 112, οι 94 απέρριψαν την πρόταση για συνεννόηση και συζήτηση μαζί σας. Ήταν ψεύδο μη κυβερνητικέ οργανώσεις, fake NGOs. Δεν εκπροσωπούν δηλαδή τον κόσμο. Πώς αυτό ε, συνδυάζεται με την απόφαση του ε, δικαστηρίου. Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό. Αισθάνομαι μεγάλη δυσφορία γιατί ανά τον κόσμο λέμε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δημοκρατία, αξίες, ανθρώπινα δικαιώματα και εδώ κάνουμε ακριβώ το αντίθετο. Οι Σαχράουι με τους ε, οποίους δεν είχατε τη δυνατότητα ή την ευκαιρία να συζητήσετε είναι στη φυλακή, γι' αυτό δεν μπορέσετε να συζητήσετε μαζί τους. Ούτε καν ξέρουν ότι υπάρχει τη συζήτηση. και βλέπω ότι για να κερδίσουμε μερικές φθηνές δωμάτες παίζουμε το βιολί των κυρίων και δεσποτών μας, με συγχωρείτε για την έκφραση. Γκουέντζιελ παρακαλώ, κυρία Μίνερ. Ευχαριστώ πρόεδρε και θα ήθελα να μου πείτε ακριβώς ε, ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι λέτε στην επιστολή της ΙΤΑ μιλάνε με σαφήνεια για την αντιμετώπιση και τη στάση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι αφορά το Μαρόκο και την Δυτική Σαχάρα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, έχει βάλει, έχει επίσης ε, αποφάσισε, αλλά αυτά τι έχει τηρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι συνάδελφοί μα είπαν ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να το δεχτούμε αυτό. Πείτε μα, λοιπόν, ε, υπάρχει μία αλλαγή πλεύσης ή μήπως είναι όλα καπνός. Μιλάτε για ευρείε διαβουλεύσει, αγαπητή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον κόσμο. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Ο κόσμο θα πρέπει να μπορεί να εκφράσει Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι θα υποστηρίξει το δικαστήριο αυτή την απόφαση ή να ζητήσουμε εκ νέου γνωμοδότηση από το δικαστήριο. Και ε, θέτω και την ερώτηση που ακούσαμε και προηγουμένω, αλλά δεν απαντήθηκε. Ερευνήσατε ποια θα είναι τα αποτελέσματα του συμφωνία ε, ε, στους ε, κατοίκους του ΡΙΦ. Και τελικά θα υπάρξει όφελος για το ΡΙΦ. Πώς θα αντιμετωπίσουμε λοιπόν και ποιον εξυπηρετούμε τελικά με αυτή τη συμφωνία. Νομίζω ότι και πάλι υποστηρίζουμε τις πολυεθνικές μας, όχι όμως τον πληθυσμό, τον κόσμο, τους πολίτες στο Μαρόκο. Ευχαριστώ από το EFTD, κυρία Μπεγκίνη. Κύριε Πεκίνη, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Όπως ξέρετε, στο παρελθόν ε, είχα αντιταχθεί και παραμένω πίστη σε αυτές μου τις πεπιθήσεις στην συμπερίληψη της γεωργίας αυτή τη συμφωνία. Ωστόσο, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν μας λέει να επανεξετάσουμε ολόκληρη τη συμφωνία, αλλά μόνο να εξασφαλίσουμε την ουδετερότητα απέναντι στους ε, Σαχράουι. Άρα παραμένει ενισχύ σε σχέση με αυτό που έχει ήδη καλύψει η συμφωνία και τις διαπραγματεύσεις που έχουν μέχρι τώρα πραγματοποιηθεί. Και το ζήτημα των Σαχράουι και η παραγωγή στη Δυτική Σαχάρα παραμένει εκρεμές λοιπόν ο ζήτημα χρειάζεται μια προς δυνατόν πιο ξεκάθαρη τοποθέτηση, ουδέτερη ενημέρωση και έχω την ίδια ε, απέτηση και από την κυβέρνηση του Μαρόκου αλλά και από του Σαχράουι. Είναι λυπηρό λοιπόν το ότι δεν είχαμε ενημέρωση πιο διεξοδική από τα όσα μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα όσα επιβεβαιώνεται κάποιες ε, οργανώσεις φαίνεται να ε, απέρριψαν την πρόταση για συνεργασία ή συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπές. Επιτροπή, άλλες δεν, δεν ε, προσεκλήθηκαν καν. Επομένως, θα ήθελα πληροφορίες για αυτές τις δύο ομάδες μη κυβερνητικών οργανώσεων. Επίσης, Υπάρχουν σαφείς ε, πληροφορίες και καταγγελίες από τους Σαχράουι ότι τα προϊόντα αυτά για τα οποία γίνεται λόγος παράγονται από ε, χωρικούς που έρχονται από το Μαρόκο εποχιακά να εργαστούν στα χωράφια για την παραγωγή της τομάτας και του πεπονιού. Ε, αυτό θα, θέλουμε, θα θέλαμε να το διευκρινίσουμε και βέβαια ξέρετε ότι για το τμήμα της Αλίας δεν είναι δυνατό να προχωρήσετε σε έγκριση χωρίς την ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προσπαθώ να καταλάβω τι προσπαθείτε να κάνετε και γιατί. Είναι ένα ζήτημα περίπλοκο, Πρόεδρε. Οπωσδήποτε περίπλοκο και δύσκολο αυτόν τον Σαχράουι δεν μπορούμε να το λύσουμε με μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Μη λησμονούμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μια συμφωνία εμπορική μόνο εδώ και για το ζήτημα των Σαχράουι μόνο, μόνη αρμόδια είναι, μόνος αρμόδιος είναι ο των Ηνωμένων Εθνών και εκεί πέρα πρέπει να λυθεί το ζήτημα. Κύριε Γκούτλαντ. Ευχαριστώ για την εισαγωγή σας. Είναι σημαντικό να πούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Είναι θέμα αρχής, πολιτικό ζήτημα, εχμής και δεν έχει σχέση μόνο με, τα, με την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο αλλά και με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο υπερητά ότι η Δυτική Σαχάρα δεν αποτελεί τμήμα του Μαρόκου και χρειάζεται συγκατάθεση του λαού προκειμένου να συμπεριληφθεί στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε μπορεί να μας εξηγήσει η Κομισιόν γιατί εστιάζεται ακόμα στα ωφέλη της, ε, στον, για τον τόπιο πληθυσμό αντί στη συγκατάθεση του λαού. Η απόφαση του δικαστηρίου ε, λέει ότι θα χρειάζεται η συγκατάθεση του λαού και ένα μεγάλο κομμάτι της επικράτειας της Δυτικής Σαχάρας δεν είναι ε, ε υποκατάληψη ε, από το Μαρόκο ενώ ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού ζει σε καταβλισμούς. Γιατί δεν ρωτώνται χωρίς τη συγκατάθεση το να συμπεριληφθεί η Δυτική Σαχάρα σε μια συμφωνία δεν είναι ουδέτερο, δεν είναι κάτι ουδέτερο. Η Κομισιόν με αυτόν τον τρόπο παίρνει θέση. Πώς περιμένετε ότι θα επηρεάσει αυτό την διαδικασία του ΟΗΕ. Ανησυχώ πάρα πολύ. Το έχω πει πανελειμμένω και με πολλούς τρόπους. Αγωνιώ. Ε, αυτό που θα γίνει θα αυξηθεί η ανασφάλεια για τις επιχειρήσεις και πιθανότατα θα δυσχερανθεί η διαδικασία έβρεσης λύσης. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την προτινόμενη συμφωνία. Ευχαριστώ. Σίλβα Περέιρο. Η ε, συμφωνία σύνδεση με το με το Μαρόκο είναι στρατηγική σημασία ε, και ταυτόχρονα όμω θα πρέπει να σεβαστούμε την διαδικασία του ΟΗΕ για, την, ε, για το καθεστώ της Σαχάρας. Καλωσορίζω τις προσπάθειες Κομισιόν που ε, επιθυμεί οι σχέσει με το Μαρόκο να ενταχθούν στο πλαίσιο της απόφασης του δικαστηρίου. Τι άλλο θα μπορούσε να έχει γίνει υπό τις παρούσες πολιτικές συνθήκες ώστε να εξασφαλιστεί μια επαρκής διαβούλευση με τον με τον πληθυσμό. Ε, έγινε αναφορά και στις επιπτώσεις της απουσίας συμφωνίας. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις ε, μιας ε, αναβολής συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν καθυστερούσαμε, αν ζητούσαμε τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις αυτής της καθυστέρησης. Ο κύριος Μαρτσελέση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, την, να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί καταφέρατε πολλά με ένα σπάρο. Συμφωνία με, για τη Δυτική Αφρική χωρίς να πατήσετε καθόλου εκεί. Αναγνωρίζετε ότι είναι μακρινή περιοχή, δεν έχετε στατιστικές, δεν έχετε αρμοδιότητες να ερευνήσετε επιτόπου. Παρ' όλα αυτά ε, ε συμφωνία από το Ραμπάτ. Μπορείτε να μου δώσετε ένα παράδειγμα παρόμοια συμφωνίας Άλλη. Δεύτερον, λέτε ότι δεν υπάρχει κυριαρχία του Μαρόκου στη Δυτική Αφρική. Παρόλα αυτά, το μεγαλύτερο κομμάτι αυτού των αρχών που, με τις οποίες διαβουλευθήκατε ε, ήταν αρχές του Μαρόκου. Ε, αυτό, από τι προκύπτει από αυτό, δεν προκύπτει ότι υπάρχει κυριαρχία του Μαρόκου. Μπορείτε να μου δώσετε ένα άλλο παράδειγμα παρόμοια συμφωνία. Τρίτον, μας λέτε ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το ρόλο ε, του με το Πολυσάριο. Και τι κάνατε με το Πολυσάριο, ε, συναντηθήκατε άτυπα, ενώ με όλους, υπάλου, με όλους υπόλοιπους ε, επισήμως. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα με το Πολυσάριο. Πιστεύετε ότι κάνοντας όλα αυτά και επιπλέον ε, στηρίζοντας de facto της, ε, το Μαρόκο, πιστεύετε ότι βοηθάτε. Τέταρτον, μιλάτε για ωφέλη στον πληθυσμό. Ποιος ε, είναι ο ιδιοκτήτης των επιχειρήσεων, των εταιριών, των βιομηχανιών αυτών ε, λοιπασμάτων. Λέτε ότι λαμβάνετε υπόψη της, ε, από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Θα μου πείτε σίγουρα ότι η νομική σα υπηρεσία έλεγξε αυτό το κείμενο και το, ε, έδωσε, ε, έδωσε, σε έδωσε το πράσινο φω. Αλλά αυτό το κάνει εδώ και 10 χρόνια. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Δεν είναι δυνατόν η Γκουε, η πράσινη και οι υπόλοιποι να μην είναι μέσα στην διαδικασία αυτή. Θα πρέπει να εκπροσωπούμαστε όλοι. Έχουμε όμω το σύστημα ΔΕΟΝ σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή ε, στι αντιπροσωπείε και αυτό γίνεται σεβαστό από όλε τι ομάδε. Ο κύριο Σόλτ. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη που άργησα. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η υπόθεση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Μόλις συζητήσαμε το θέμα της Μολδαβία. γιατί είναι σαφές ότι όλες οι προϋποθέσεις για την παροχή μακροοικονομικής αρρωγής δεν πληρούνται, παραβιάζονται διαρκώς. Μιλάμε για την ευθύνη του συνομοθέτη σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση της διαδικασίας και αυτό σε ό,τι αφορά και τις ερωτήσεις για τη Βετική Σαχάρα. Εξ όσων κατανοώ, πολλές ερωτήσεις ε, με βρίσκουν σύμφωνο. Το βασικό πρόβλημα θεωρώ βρίσκεται στο εξή σημείο. Γιατί δεν μιλάμε στη Βυτική Σαχάρα με τον κόσμο. Γιατί δεν ανήκει στο Μαρόκο. Αυτό είναι το διεθνέ δίκαιο. Και αυτό το τονίζει διαρκώς. Ε, το τονίζουν διαρκώς οι εκπρόσωποι του ΟΗΕ. Γιατί λοιπόν δεν το κάνουμε αυτό. Γιατί δεν το κάνετε εσείς αυτό. Δεύτερη ερώτηση. Γιατί επιμένετε για να υπάρξει όχι μία συμφωνία μόνο για το Μαρόκο όπως ε, συνήψαν οι ΙΠΑ. Γιατί δεν είναι δυνατόν αυτό. Πώς θέλετε να γίνει διάκριση, γιατί όλες οι άλλες διαδικασίες ε, παρακολούθησης follow-up είναι πολύ πιο περιπλοκές. Ποιος θα καθορίσει, ποιος προέρχεται από πού. Θα περιοριστώ λοιπόν στι δύο αυτέ ερωτήσει, γιατί νομίζω ότι έχουμε κάποια κρίσιμα σημεία τα οποία θα πρέπει να μα απασχολήσουν για να κατανοήσουμε ακριβώ ε, και να συνοηθούμε μεταξύ επιτροπή και Συνομοθέτη. Ευχαριστώ. Από πλευρά μου έχω να σα ρωτήσω ποιο είναι το καθεστώ ε, τη μελλοντική ε, αγορά στην Αλία. Δεν είμαστε Επιτροπή Ελία, αλλά θεωρώ ότι από θεσμική άποψη και από συνταγματική άποψη υπάρχει σύνδεσμο. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι δύο συμφωνίες εκ παραλληλού. Πώς έχουν λοιπόν τα πράγματα. Τέντσλερ και Πικέ. Για πέντε λεπτά ο καθένας. Okay. Uh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Πολλές ερωτήσεις. και δεν είμαι βέβαιη ότι με το λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας θα μπορέσω να απαντήσω σε όλε εξ αυτών, αλλά είναι και πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε τη συζήτηση και φυσικά είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε και διμερώς. Ετέθησε το ερώτημα των διαβουλέσεων και του πληθυσμού. Τι σημαίνει πληθυσμός, τι σημαίνει κόσμος, τι σημαίνει λαός Volk στα γερμανικά. Αυτά θα τα απαντήσει ο συνάδελφο από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Για να απαντήσω σε ένα σχόλιο το οποίο έγινε. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν προνομιακές, ε, προνομιακοί δασμοί. Όπως είπε ο συνάδελφός σας λοιπόν, αν δεν ε, αναλάβουμε δράση, αν δεν δώσουμε προνομιακό καθεστώς τώρα, ουσιαστικά τιμωρούμε τον κόσμο στη Δυτική Σαχάρα, τότε μπορούμε με υψηλότερους δασμούς. Και επιδεινώνουμε το επενδυτικό κλίμα και το επιχειρηματικό κλίμα. Για το ερώτημα του κατά πόσον θα μπορούσαμε να κάνουμε μία όχι εφάπαξ διαβούλευση όπως γίνεται τώρα, αλλά να δημιουργηθεί μια διαρκής διαδικασία διεξαγωγής διαβουλεύσεων. Το είπα εισαγωγικά νομίζω ότι θα ήμασταν δεδομένοι και είχαμε ζητήσει από τους μαροκινούς ομολόγους να ξεκινήσουν μια διαδικασία παρακολούθησης διαρκούς ανταλλαγή. τουλάχιστον άπαξ ετησίως για να υπάρχει ανταλλαγή για να δούμε κατά πόσον η συμφωνία πραγματικά έχει το αποτέλεσμα το οποίο επιθυμούμε ή κατά πόσον χρήζει βελτίωσης και θα πρέπει λοιπόν αυτό να ληφθεί υπόψη για να ληφθούν υπόψη ναι, και ε, οποιασδήποτε εξελίξει στα πλαίσια της Eurolab. Για την γνωμοδότηση από πλευράς του δικαστηρίου. Να καλέσω τους αξιότιμους βουλευτές να αναλογιστούν και την πολιτική τους ευθύνη και την νομική τους ευθύνη. Νομίζω ότι εδώ μιλάμε για την πολιτική ευθύνη της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπό την έννοια αυτή, το Κοινοβούλιο ενδεχομένω να θέλει το λάδι αυτό υπόψη. Οι συνέπειε μια καθυστέρηση, ε, το ανέφερα ήδη. Οι συνέπειε μια καθυστέρηση ε, θα ήταν ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει προνομιακό καθεστώ. Τέλος. για τη συμφωνία για την αλληλεία να απαντήσει ο κύριος Πικέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχάς, για τις διαβουλεύσεις, την μέθοδο που ακολουθείτε και την επιλογή συνομιλητών. Να τονίσω καταρχάς ότι η δικαστική απόφαση δεν διευκρινίζει τίποτε για το πώς θα πρέπει να διοργανωθούν οι διαβλέψεις. Δεν ε, αναφέρει τίποτε τέτοιο ούτε στη Συμφωνία για την Αλία, ούτε στην Συμφωνία για τη Γεωργία. Άρα αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου ως Ευρωπαϊκή Υπηρεσία και ως Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να ερμηνεύσουμε το πώς θα προχωρήσουμε σε ένα πολύ περίπλοκο θεσμικό υπόβαθρο. Τι επιλέξαμε. Να μην έχουμε ένα καθεστώς προνομιακής μεταχείρισης ε, των συνομιλητών μας. Αποφασίσαμε να μην ε, συζητήσουμε μόνο την κυβέρνηση του Μαρόκου ή του Πολυσάριο. Και τους δύο. Θέλαμε να υπάρχει μια πολύ ευρύ, ομάδα συνομιλητών και ε, δυστυχώς μετά από επανελειμμένες απόπειρες κανείς δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Έτσι έχουν τα πράγματα το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων παρόλα αυτά. Είναι αξιόπιστο. Πρόκειται για μια αξιόπιστη ομάδα συνομιλητών, ε, την οποία έχουμε πλέον ενώπιόν μας. Είναι πραγματικοί άνθρωποι, πραγματικές ε, οργανώσεις, πραγματικές ΜΚΟ. Εγώ ο ίδιος έκανα τις συνομιλίες αυτές και σας το λέω από πρώτο χέρι. Σε ό,τι αφορά το στοιχείο αυτό λοιπόν των διαβουλεύσεων. το ερώτημα του γιατί δεν στραφήκαμε και δεν πήγαμε οι ίδιοι στη Βυτική Σαχάρα. Οι συνομιλίες αυτές θα να γίνουν σε ένα περιβάλλον με την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία όπου ο κόσμος θα μπορούσε να εκφέρει την άποψή του. Και αυτό για παράδειγμα προβλέπετε για τον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων και των διαβουλεύσεων, για παράδειγμα, στην Δυτική Σαχάρα σε ό,τι αφορά την Αλία. Τώρα, το ερώτημα του Προέδρου για την ε, Συμφωνία για την Αλία. Συνεχίζονται οι συζητήσει, έχει δοθεί εντολή τον Απρίλιο από πλευρά του Συμβουλίου. Συνεχίζονται λοιπόν ε, οι συνομιλίε και για μια εντελώ καινούργια συμφωνία για την Αλία, αλλά και για τι συγκεκριμένε πτυχέ, τεχνικέ δηλαδή πτυχέ του πρωτοκόλου σε ό,τι αφορά την ποσότητα των αλευμάτων, των χρημάτων που χρησιμοποιούνται και την πολιτική πολιτικής διάστασης, όπως για την συμφωνία για τα γεωργικά, για τα αγροτικά προϊόντα. Θα είναι λοιπόν ένα ευρύτατο πακέτο το οποίο είναι υποδιαπραγμάτευση. Δεν μπορώ να σας δώσω ένα σαφές ε, χρονοδιάγραμμα, αλλά πραγματικά προσπαθούμε να κινηθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Λελόντ, για να ολοκληρώσουμε. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Απλώς για την αυτοψία, ε, την αποστολή αυτή που θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να γίνει στη Δυτική Ζαχάρη, εξ αρχής το έχω υποστηρίξει. Αρέσει δεν αρέσει τους ε, Μαροκινούς, πρέπει να πάμε. να κάνουμε το, τα πάντα για να λάβει χώρα αρχές Σεπτεμβρίου το θέμα, η επίσκεψη αυτή και νομίζω ότι η διαδικασία είναι γνωστή. Bah, écoutez, euh, on va voir comment ça se passe, mais on va faire en sorte que ça. Excusez-moi, je pense qu'on peut faire un effort. Enfin, voilà. Et... Τα σχόλια ήταν εκτός μικροφώνου. Και βεβαίως θα πρέπει να κάνουμε όσο, να παρακολουθήσουμε όσο δυνατόν πιο προσεκτικά τα όσα κάνει ο κύριο Κόλλος και βεβαίως να παρακολουθούμε το ε, χρονοδιάγραμμά του. Τον Οκτώβριο νομίζω έπρεπε προβλέπεται να καταθέσει την έκθεσή του, επομένως ας, την, ας παρακολουθήσουμε, έπρεπε ήδη να είχαμε ε, παρακολουθήσει το πρόγραμμα του πιο στενά. Κλείσαμε, λέει ο Πρόεδρος, το 24, το 25 στα διάφορα όχι. Τι ωραία. Το ωραιότερο κομμάτι, λέει ο πρόεδρος τη ημερησία διάταξη, το 26. Προσεχή συνεδρίαση 9 και 10 Ιουλίου. Και αυτά. Σας ευχαριστούμε και επισημαίνουμε στις ερμηνείς ότι τελειώσαμε στην ώρα μας.